Okay, we'll get started. You Γεια σας, έχετε το σχέδιο ρίσκιας διάταξης. Ε, φαντάζομαι ότι το δέχεστε. Μπορούμε να την εγκρίνουμε λοιπόν την μερίσια διάταξη. Εάν συμφωνείτε να περάσουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο τη διάταξη, το σημείο 2, παρουσίαση από την ΓΔ Κλίμα της πρότασης για το πρόγραμμα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών στην πολιτική αεροπορία. Κυρία Μπάντραμ εδώ. Ελίνα Μπάντραμ. Μάλιστα. Βλέπετε ότι υπάρχει αθρότατη προσέλευση δεν ήθελα να έχουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας μόνο την Πέμπτο πρωί, αλλά δεν φαίνεται ότι έχω πείσει μέχρι τώρα τις υπηρεσίες της, ε, του Κοινοβουλίου. Τέλος πάντων έτσι έχουν τα πράγματα, αυτό το ηλίθιο σύστημα, αυτά μας επιβάλλει. Λοιπόν, έχετε το λόγο. Okay, thank you. Good morning. And I have... Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα προνόμιο ε, το θεώρησα που με βάλατε πρώτη-πρώτη την πέμπτη το πρωί. Πολύ έτσι καλό σλότ. Okay. Um, indeed. Uh, as you know... Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια πρόταση για τροποποίηση ε, του συστήματος εμπορίας και μετών εκπομπών για την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 16 Οκτωβρίου και αυτό έρχεται σε απάντηση στο ψήφισμα της συνέλευσης της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας. Ε, συμφωνήθηκε στις 4 Οκτωβρίου συγκεκριμένα. Και σε αυτό το ψήφισμα η ΔΟΠΑ αναφέρει, σημειώνει τις επιστημονικές απόψεις ότι αφορά τις μειώσει εκπομπών, θεωρεί ότι είναι αναγκαίες. Συμφωνεί να συμβάλλει ε, στο να υπάρξει συμβολή και από τον τομέα της ε, πολιτικής αεροπορίας. Ίσως θα θέλατε να ξέρετε ότι εκπομπές από την πολιτική αεροπορία φαίνεται ότι θα αυξηθούν ε, κατά 500-800% μέχρι το 2050 από τα επίπεδα του 2005 και γι' αυτό οι εκπομπές αεροπορίας περιλαμβάνονται στις πολιτικές ε, της Ένωσης για τις εκπομπές και ιδίως ό,τι αυτό το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Ποια είναι η ε, εικόνα της βιομηχανίας. Ε, ξέρετε ότι η ΙΑΤΑ στην ετήσια γενική της συνέλευση του Ιουνίου φέτος ενέκρινε ένα ψήφισμα που επίσης αναγνωρίζει την ανάγκη μέτρων ε, αγορακεντρικών βασισμένων στην αγορά και την εκπόνηση ενός οδικού χάρτη για την εκπόνηση των μέτρων αυτών από το 2020 και μετά θεωρούν τις προβολές τους ότι θα είναι απαραίτητα αυτά τα μέτρα για να εκπληρωθούν οι στόχοι της ΔΟΠΑ αλλά και οι στόχοι της αγοράς. Θα δείτε ε, από αυτές τις προβολές ότι υπάρχει μια φιλόδοξη υπόθεση, σενάρια ότι θα υπάρξουν ε, ε, νέες τεχνολογίες που πριν το 2050 θα έχουν ανακαλυφθεί νέες φιλοπεριβαλλοντικές τεχνολογίες που θα συμβάλλουν τα μάλλα στη μείωση των εκπομπών. Είναι βέβαια φιλόδοξο το σενάριο αυτό. Πάντως προς το παρόν θεωρείται ότι απαιτούνται ε, αυτά τα κεντρικά μέτρα. Τι καλύπτουμε αυτή τη στιγμή. Καλύπτουμε όλες τις διαδρομές, όλα τα δρομολόγια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΟΧ ε, και επίσης τα αεροδρόμια τρίτων χωρών. Τις αφήξει εκεί. Έχουμε το γεωγραφικό πεδίο από την οδηγία του 2008. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφαθεί ότι συνάδει πλήρως και με τη Σύμβαση του Σικάγου και με τις άλλες διατάξεις προσέγγισή μας. Σε ό,τι αφορά τώρα το εφιστάμενο δίκαιο, εμείς πάντοτε ήμασταν της άποψης ότι οι πολυμερείς ε, ε, μηχανισμοί, οι πολυμερείς διαδικασίες είναι ένα κομβικό σημείο και περιμέναμε να έχουμε ένα αποτέλεσμα ώστε να μπορέσουμε την προσέγγιση μας ε, της ΕΔΕ να την ε, ευθυγραμμίσουμε στη γενική, στην παγκόσμια προσέγγιση. Τι έγινε λοιπόν, στην Γενική Συνέλευση της ΔΟΠΑ τον Οκτώβριο το 2013. Υπήρξε μια σαφής απόφαση να σχεδιαστεί αυτό το μέτρο, το παγκόσμιο το αγορακεντρικό market-based measure που θα εφαρμόζεται από το 2020 και μετά. Η απόφαση θα ληφθεί το 2016. Ε, λίγο λυπηρό ήταν το γεγονός ότι δεν σημειώθηκε πρόοδος σε ό,τι αφορά το πλαίσιο περιφερικής δράσης και στα πλαίσια της περιφερικής δράσης μάλιστα Από το ψήσιμο το 2010 επελέγει μια διατύπωση που αφορά τις διαπραγματεύσεις και τις διαβουλεύσεις σε περίπτωση υλοποίησης διάμεσων αγροκεντρικών μέτρων. Ένα άλλο σκέλος της παραγράφου έχει να κάνει με τον κανόνα των ελαχίστων, όπως τον λέμε, στην περίπτωση περιφερειακών μέτρων ώστε τα δρομολόγια από και προς αναπτυσσόμενα κράτη με λιγότερο από το 100% μερίδιο πολιτικής έργου, θα εξαιρούνται στο πλαίσιο των ενδιάμεσων αυτών ε, μέτρων. Ποια είναι η δική μας ε, απάντηση. Όπως σας είπα, εστιάζουμε τις προσπάθειες μας σε μεγάλο βαθμό σε μια παγκόσμια αυτή διαδικασία. Έχουμε επενδύσει τεχνικές ομάδες εργασίας που επεξεργάζονται παγκόσμια μέτρα. Θα συνεχίσουμε το έργο αυτό σε όλη τη διάρκεια του περσινού ε, τους και στους τελευταίους 18 μήνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη της Ένωσης συμμετείχαν ενεργά στο έργο των τεχνικών εμπειρογνωμόνων ε, ώστε να τους βοηθήσουν να ε, προσδιορίσουν και το μοτίβο και τη μορφή αυτών των παγκοσμίων. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και η πρόθεσή μας είναι ένα μεγάλο φάσμα ε, εμπλεκομένων από τον ακαδημαϊκό ερευνητικό κόσμο και από την κοινότητα πολιτών να συμμετάσχουν σε αυτές τις προσπάθειες ώστε να έχουμε την εκτελεστική απόφαση μέχρι το 2016 και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με τη γενική την παγκόσμια αυτή προσέγγιση. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η Τυλιβία λήθος ε, σε αυτό το μέτρο θα είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καν συμφωνήσει ε, για όλα τα συστατικά ε, που θα απαρτίζουν, θα σε αποτελούν αυτό το, αυτά τα μέτρα. Πρέπει να γίνει λοιπόν προσπάθεια σε αυτήν την κατεύθυνση. Ένα άλλο σκέλος της απάντησής μας είναι η πρότασή μας. Τι προτείνουμε λοιπόν. Έχουμε καταθέσει μια πρόταση που περιορίζει το στόχο της, ε, του συστήματος ε, δικαιωμάτων ε, εμπορίε δικαιωμάτων εκπομπών για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος. Για το έτος αυτό, το 2013, για τις εκπομπές, έχουμε αυτή τη λεγόμενη μεταβατική φάση, ώστε να κάνουμε την τεχνική προπαρασκευή και για φέτος καλύπτουμε μόνο στην πρότασή μα τη κυκλοφορία μεταξύ αεροπορίων του ΕΟΧ με βάση την απόσταση, τη διανηθής απόσταση. Όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι προετοιμασίε και θα ε, είμαστε σε θέση να σας ε, δώσουμε την ε, νομική βάση και να την κοινοποιήσουμε και στους αερομεταφορείς, θα έχουμε μια προσέγγιση τότε η οποία θα καλύπτει την ενδοκοινοτική, ε, τις μεταφορές οι τρίτες χώρες, η κίνηση μεταξύ τρίτων χωρών θα καλύπτεται μόνο σε ό,τι αφορά την απόσταση που διανύεται εντός ε, του χώρου, του χώρου Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΟΧ. Θα δούμε και την εξοεδαφικότητα. Υπάρχουν κάποιες αξιώσεις, ε, τα έχουμε συζητήσει και τα έχουμε δει τα τελευταία τρία χρόνια. Θα τα αντιμετωπίσουμε τα σχετικά θέματα. Τους κανόνες των ελαχίστων του ψηφίσματος ε, του, της ΔΟΠΑ του έχουμε συμπεριλάβει. ποια δρομολόγια θα εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογή. Η πρότασή μας ε, είναι περιορισμένη χρονικά και σχετίζεται, συνδέεται και με την όλη διαδικασία στο πλαίσιο της ΔΟΠΑ. Βλέπετε εδώ τι καλύπτουμε, τις πτήσεις εντός ΕΟΧΑ, πλήρης ε, κάλυψη όλων των αποστάσεων, δηλαδή αεροδρόμια τα οποία είναι εντός χωρών μελών του ΕΟΧ και αεροδρόμια που βρίσκονται και στις από απόκεντρες περιφέρειες του ΕΟΧ. Εδώ βλέπετε την κάλυψη των πτήσεων σε σύγκριση με την υφιστάμενη οδηγία. Είδατε το σχέδιο που έχουν την πλήρη κάλυψη πριν. Με αυτή την πρόταση τώρα που διατυπώνουμε θα καλύπτουμε από το London Heathrow για παράδειγμα στο Σαν Φρανσίσκο μόνο το 8,7% τις εκπομπές που αυστηρά εκπέμπονται, γίνονται εντός ε, του περιφερειακού εναέρου χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξαιρείται η ε, διαδρομή πάνω από τον Ατλαντικό, πάνω από τον Καναδά, πάνω από τις ΗΠΑ. Αυτό είναι ένα άλλο γράφημα για να δείτε ακριβώς τι θα ισχύει όταν βγει ε, τον Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ενέριο Χώρο το αεροπλάνο δεν καλύπτεται πλέον, ε, δεν καλύπτεται εκπομπέ του. Αυτό είναι μια, ένα συνδυασμός ε, των διαφόρων παραδειγμάτων κάλυψης που προτείνονται. Για την Ισλανδία βλέπετε, επειδή η απόσταση πάνω από τα διεθνή ύδατα την ε, ανοιχτή θάλασσα. Βλέπετε ότι περιλαμβάνεται ένα κομμάτι του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Χώρου, έχουμε και την Νορβηγία. Καλύπτεται μέχρι τα 12 μίλια από την ακτή της Ισλανδίας. Δεν καλύπτεται όμως άπαξ και βγει από τα 12 ναυτικά μίλια ε, της Ισλανδίας στο αεροπλάνο. Θα υπάρξει μια αλλαγή επίσης στην παρακολούθηση, ε, την υποβολή αναφορών και την επαλήθευση στο MRV. Έχουμε κατ' εξαίρεση ένα κύκλο δύο ετών, ε, κύκλο συμμόρφωσης δύο ετών, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν ε, οι αερομεταφορείς για το νέο καθεστώς. Αυτό το προτείνουμε για το 2013-2014, να γίνουν απαραίτητοι υπολογισμοί και να καλύψουμε, να κάνουμε και τις προτάσεις μας για την κάλυψη ε, των δρομολόγων προς τρίτες χώρες. Δύο είναι οι προτάσεις ε, για τις πτήσεις ε, από τρίτες χώρες, να ισχύσει το τρέχον σύστημα Μαρβή ή να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις από το Eurocontrol στο τεφρά τις εκπομπές. Δηλαδή πόσες εκπομπές εξωτερικού του άνθρακα εκπέμπονται εντό του περιφερειακού ενέργου και μετά έχουμε ένα πολλαπλασιαστή που ισχύει. Νέες εξαιρέσεις που προτείνονται τώρα για μικρούς ε, εκπομπούς ας πούμε, αυτούς που εκπέμπουν λίγους, δηλαδή εκπομπές κάτω από χίλιους τόνους διοξιδίου. Βλέπουμε ότι έχουμε μία μείωση που δεν φτάνει καν τη μία ποσοστία μονάδα, 0,2% ε, στην κάλυψη 2.200 ε, φορείς δεν θα καλύπτονται πλέον, τεράστια ε, μείωση του διοικητικού άχθους των αρμόδιων αρχών και των φορέων γενικώ. Επίσης προτείνουμε απλουστευμένες διαδικασίες για όσοι εκπέμπουν λιγότερο από 25.000 τόνους δεξιδιού άνθρακα το χρόνο για να μπορούν να χρησιμοποιούν έναν απλουστευμένο μηχανισμό ε, του Eurocontrol. Θα υπάρχουν ε, επίσης γραμμικές μηχανικές προσαρμογές για τον πληστηριασμό και για τα ελεύθερα δικαιώματα εκπομπών. Η ποσότητα των ε, δικαιωμάτων αυτών θα μειωθεί κατά αναλογία με τη νέα κάλυψη. Η κυκλοφορία ε, από τρίτες χώρες θα καλύπτεται μόνο για τη διαδρομή εντός του περιφερειακού εναέριου χώρου της Ένωσης. Αυτά είναι λοιπόν τα σημερινά στοιχεία. Μέχρι στιγμή έχουμε πλήρη κάλυψη της κυκλοφορίας από τρίτε χώρες. Στο εφιστάμενο δίκαιο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια ομαλή διαδικασία συναπόφασης για να φτάσουμε σε μια βιώσιμη ζώνη προς, ε, βιώσεων ε, σύντομα. Θα πρέπει μέχρι τον Απρίλιο 2014, είναι το λεγόμενο surrender deadline αυτό, πρέπει να έχουμε αποφασίσει. Οπότε θα είναι άκρος χρήσιμο για όλους μας να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε επί μιας πρότασης και μιας νομικής προσέγγισης που θα μας δώσει τη δυνατότητα να τη μεταφέρουμε ε, την απόφαση αυτή στους ε, μεταφορείς μας αλλά και σε τρίτους, ε, σε φορές από τρίτες χώρες. Τρει μήνε τουλάχιστον απαιτούνται για τη μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο, μετά δηλαδή από την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και η πρώτη προθεσμία, η νέα προθεσμία συμμόρφωση, θα είναι οι αρχέ του 2015, ώστε να δοθεί απαραίτητο χρόνο για να γίνουν οι απαιτούμενε τροποποιήσει στο καθεστώ συμμόρφωση και στι πρακτικέ ε, υποβολή αναφορών. Ολοκληρώνω με αυτά και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ε, με τα χαράς να απαντήσω σε ερωτήσεις σας. Thank you very much, Mr. Gross. Ο κύριος Γκρός. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και εξήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολλά έχουμε, βέβαια, να επισημάνουμε. Θα είναι όμως αναγκαίο να επικεντρωθώ σε κάποια ορισμένα σημεία μόνο. Άρα θα πω ότι σε διεθνέ επίπεδο δεν φαίνεται να έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο η δράση και οι επιλογέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονό ότι μέσα σε τρία χρόνια, τρει φορέ σχεδόν, χρειάστηκε να αλλάξει αυτή η βάση, δεν μα βελτιώνει την αξιοπιστία μα. Εξού και θεωρώ πως διδασκόμενοι από το παρελθόν θα πρέπει να διαμορφώσουμε διαφορετικές προοπτικές για το μέλλον. Δύο ερωτήσεις λοιπόν, διότι καταπλήσουμε για το ότι τα κράτη τα οποία δεν ε, επηρεάζονται καν από τις δικές μας ε, δράσεις, τα μέτρα μας, ε, εντυπωσιάζουμε λοιπόν για τα κράτη αυτά έχουν ενωθεί κατά των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουν δημιουργήσει αυτό το μέτωπο αντίστασης. Δεύτερον, το σύστημα φέρνει, ε, συνεπιφέρει και κάποιες υποχρεώσεις. Και θα ήθελα να ξέρω αν είμαστε σε θέση να τιμήσουμε αυτές τις υποχρεώσεις ή εάν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Για το μέλλον θα ήθελα, να είμαι να ακούσω από τους συναδέλφους ε, οι πολιτικές τους ομάδες πώς βλέπουν την κατάσταση γιατί νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να προετοιμάσουμε μια μεταβατική φάση μέχρι το 2016 με ευελιξία. η οποία θα μας επιτρέπει και να διαφυλάξουμε την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της ΑΕΚΕΟ και να προετοιμάσουμε την ε, μεταγενέστερη φάση και να δεχθούμε βέβαια από το παρελθόν μας. Αλλά επίσης θα έλεγα ότι υπάρχει και μια άλλη επιλογή. Να μην προετοιμάσουμε τώρα μια μεταβατική φάση, αλλά να πούμε από τώρα, από το 16 και μετά τι θα ισχύει, για να είμαστε πιο προσεκτικά προετοιμασμένοι. Και να περιμένουμε να έχουμε ορίσει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και όχι ένα προσωρινό. Επίσης, βλέπω ότι έχουν ζητηθεί ε, γνωμοδοτήσεις πολύ άριθμες για την ποιότητα και το αποτελέσματα των διαφορών ε, αποφάσεων, αλλά όταν ε, μιλάμε για πολιτική αεροπορία, οι συνθήκες του Σικάγου είναι αυτές οι οποίες επικρατούν και άλλωστε εξαρτώμεθα και από τις επιλογές και άλλων κρατών που είναι μέλη της ΕΚΑΟ. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να λάβουμε αποφάσεις οι οποίες θα έχουν και αποτελέσματα και μια, ε, θα έχουν έναν ορίζοντα χρονικό μεγάλο. Επίσης, ε, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και το θέμα των διμερών συνθήκων ή συμβάσεων θα μπορούσαμε να συνάψουμε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων κρατών, μεγάλων εταίρων όπως οι ΗΠΑ ή άλλες περιφέρειες του κόσμου. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση εναλλακτική σε σχέση με τις διεθνείς συμφωνίες. Γι' αυτό καλό θα ήταν να εξετάσουμε τι είδους δυνατότητες μπορεί να μας προσφέρουν τέτοιου είδους διμερείς συμφωνίες. Και τέλει, ελπίζω να μην ε, αφήσουμε να περάσει ο χρόνος περιμένοντας τι θα γίνει μετά το 2016, αλλά ήδη να σχεδιάσουμε το 2020. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλκαντράουι. Ευχαριστούμε πολύ την ε, Κομισιόν για την παρουσίαση που έκανε. Ευχαριστούμε πολύ και τον συνάδελφο Γκρόσου ε, που είναι εισηγητής. Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Μια πρώτη παρατήρηση λοιπόν για να πω ότι ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως δείξαμε υπερβολική αισιοδοξία ή μάλλον φιλοδοξία ε, στην διατύπωση της νομοθεσίας μας και η απεσιόδοξη πούν ότι τώρα οπισθοδρομούμε ε, ή ότι θα πρέπει να οπισθοδρομήσουμε η εφαρμογή των κανόνων σε διεθνές επίπεδο θα είναι κάτι πιο δύσκολο Βεβαίως, οι αισιόδοξοι μπορούν πάντα να πούν ότι ναι, μεν είχαμε πολύ φιλόδοξη νομοθεσία, αλλά παρόλα αυτά οθήσαμε τα πράγματα προς τα εμπρός. Βεβαίως, όλα θα εξαρτηθούν από τις προόδους που θα καταγραφούν στο μέλλον κυρίως δε το τι θα γίνει ε, με την σημαντική ε, προθεσμία του 2016. Εκεί θα δούμε ποια τροπή θα πάρουν τα πράγματα. Ε, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας ε, φαίνεται ότι τα πράγματα τα έχουμε δει σωστά, αλλά μονούμε την πολιτική διάσταση του ζητήματος. Ε, και βεβαίως πολλά μέτρα μπορούν να ληφθούν κατά, των ευρωπαϊκών, κατά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και μπορεί να καταλήξουμε σε έναν εμπορικό πόλεμο. Η πρόταση που βρίσκεται τώρα μπροστά μας νομίζω ότι μοιάζει ανησυχητικά ε, στην πρόταση που είχε φτάσει στην Επιτροπή Μεταφορών πριν από μερικά χρόνια για στην ουσία ευρωπαϊκή διάσταση ε, και αντιμετώπιση, κανόνες ευρωπαϊκούς που δεν θα ακολουθούνται σε διεθνές επίπεδο. Θα δούμε τι θα γίνει και στη μεταβατική περίοδο, αλλά έχω την αίσθηση πάντως ότι κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δύο ερωτήσεις ενδεχομένως να θέσω στην, στην ε, Κομισιόν. Πρώτον, μέχρι ποιο βαθμό έχει μελετηθεί ο αντίκτυπος των μέτρων αυτών στη δικιά μας ε, αεροπορική βιομηχανία ε, και ποια θα είναι τα, ποιος θα είναι ο άμεσος αντίκτυπος μετά την εφαρμογή. Εννοώ το εξής υπάρχει κίνδυνος να δημιουργηθούν hub εκτός των κόμβι, εκτός ε, της ε, ενωσιακής ε, επικράτειας. Κυρίως προς τη Μέση Ανατολή και αυτό θα παρουσιάζει το πλεονέκτημα να μην υπόκειται στους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αυτό θα έχει αντίκτυπο λοιπόν στη δικιά μας αεροπορική βιομηχανία. Το έχετε μελετήσει αυτό. Δεύτερον, κάτι που δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Για τις πτήσεις οι οποίες ε, περνούν πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς προσγείωση επί του ενωσιακού εδάφους. Εκεί εφαρμόζεται ο ενωσιακός κανόνας. Επίσης, να συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που είπε ο Μάθιου Γκρόσο όσον αφορά τις τρίτες χώρες. Πιστεύω ότι είναι απολύτως ουσιώδες οι ε, συμφωνίες οι οποίες ε, τίθενται υπό διαπραγμάτευση ε, τούτη την εποχή θα πρέπει να λάβουν υπόψη και τα ζητήματα της αεροπορίας. Αυτά τα ζητήματα θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να τα συζητάμε έτσι ώστε ενδεχομένως να καταλήξουμε ε, σε ε, συμφωνίες ε, διμερείς, έτσι ώστε να ενισχύσουμε τη διαπραγματική μας θέση, έτσι ώστε να επιτύχουμε μια σύμπραξη. Ευχαριστώ κύριε Μάιστερ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ την Επιτροπή για την έκθεσή της. Είναι μια δύσκολη απόπειρα αυτή στην οποία αποδιόμαστε. Σε άλλε ε, περιπτώσεις έχουμε ήδη αποτύχει. Ίσως τώρα πρέπει να κάνουμε μια ακόμα προσπάθεια για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία για το ε, διοξείδιο του άνθρακα σε επίπεδο ΙΚΑΟ και μέχρι το 2016 έως και το 2020 για να έχουμε τότε μια σαφή απάντηση. Θα συμφωνήσω σε πολλά από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι πριν από μένα. Πρέπει να κοιτάξουμε με ανοιχτό πνεύμα όλη αυτή την υπόθεση, αλλά επίσης ε, οποιαδήποτε απόφαση και αν λάβουμε με μέλημα το περιβάλλον και την προστασία από την κλιματική αλλαγή κτλ. δεν πρέπει να λησμονούμε ότι βλάπτουμε, παραβλάπτουμε την ε, πολιτική μας αεροπορία, την, την ευρωπαϊκή πολιτική αεροπορία. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι σκοπός μας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει εμείς οι Ευρωπαίοι να βρούμε μια λύση η οποία ναι βεβαίω θα είναι λογική ω προς το περιβάλλον αλλά δεν θα επηρεάζει σοβαρά και τις ε, ε, πολιτικές, ε, δεν θα επηρεάζει και την επιβίωση της πολιτικής αεροπορίας. Πρέπει λίγο πολύ να τετραγωνίσουμε τον κύκλο, όπως θα έλεγα, αλλά ε, επαναλαμβάνω, ναι, να προστατεύσουμε το περιβάλλον, χωρίς όμως να κινδυνεύσει η πολιτική αεροπορία. Και μπορούμε να έχουμε ένα δικό μας σύστημα, ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο μπορούμε να προωθήσουμε και μέσω των διμερών μας συμβάσεων και όχι μόνο μέσω νέων συμφωνιών στις οποίες θα επιδιώξουμε να συνάψουμε αλλά να το εντάξουμε μέσα σε υφιστάμενες συμφωνίες Φερρυπίν με τον Καναδά έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία και πολύ καλές σχέσεις και θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε και, να προετοι... και προετοιμάζοντας το 2016 να διαμορφώσουμε για την Ευρώπη ρεαλιστικά δεδομένα ασκώντας και πίεση προς την ε, ΙΚΑΟ λέγοντας ότι ναι, μπορεί δύο φορές ε, να αποτύχαμε, αλλά δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Αυτά είναι ολίγης. Κρέμερ. Κύριος Κρέμερ. Ναι, τόντι πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρώπη να καταβάλει προσπάθειες ε, και να επιδιώξει λύση σε παγκόσμιο επίπεδο. Είχαμε προσφύγει Χάσαμε νομικά, πολιτικά δεν υπήρχαν επιχειρήματα και γιατί το λέω αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι ήττα, διότι δεν υπόθηκε τίποτε το συγκεκριμένο. Δηλαδή το μόνο που γίνεται είναι να ξανασυζητάμε και να λέμε το 2000 16, το 2013, το 2010, το 2001 τα ίδια ακριβώς πράγματα. Γιατί, διότι δεν υπήρχε εναλλακτικό σχέδιο, δεν υπήρχε επαρκή προετοιμασία. Οι αεροπορικές εταιρείες ε, στη Γερμανία, για να σας εξηγήσω, έχουν αποδεχθεί το σύστημα μείωσης των εκπομπών μόνο και μόνο για να αποφύγουν την, ε, το, την επιπλέον επιβάρυνση από την κυροζήνη, γιατί ήταν τόσο ακριβή η κυροζήνη που τους ερχόταν πιο συμφέρουσα η επιλογή του συστήματος ανταλλαγών εκπομπών. Ε, λοιπόν, εφόσον έχουμε ε, αποτύχει στο επίπεδο αυτό θα χάσουμε ταυτόχρονα και τον φόρο από την κυροζήνη, τα 16 αυτά δισεκατομμύρια που αντιστοιχούν στον φόρο από την για την κυροζήνη καλύτερα σε όλες τις αεροπορικές μεταφορές στην Ευρώπη. Και ναι, ε, μπορεί να έχουμε περισσότερε αεροπορικές μεταφορές, περισσότερη πυκνότητα κυκλοφορίας στον αέρα, αλλά δεν πρέπει να λησμονούμε και τις αρνητικές επιπτώσεις και το κόστος που αυτές συνεπιφέρουν. Και όταν έχουμε μία πτήση η οποία φεύγει από την Ευρώπη για να πάει μέχρι τις Ηνωμένε Πολιτείες, με μετεπιβίβαση, πριν από τη Γερμανία στην Πορτογαλία και από την Πορτογαλία στις Ηνωμένε Πολιτείε, τότε υπάρχει επιβάρυνση από την κυροζήνη με το φόρο ε, της ε, έτσι λοιπόν ε, ο επιβάτης ο οποίος θα πάρει ένα εισιτήριο με επιβάρυνση 30 ευρώ για το φόρο της κυροζήνης δεν θα καταλάβει τη διαφορά και δεν θα διστάσει να πάρει τον, την πτήση με την επιβίβαση. Οι δε άλλοι οι οποίοι πάνε απευθείας περνάνε από τη ε, Σιβηρία και πληρώνουν το σχετικό τέλος. Ε, Επομένω, θα μπορούσαμε και εμεί να κάνουμε ωραιότατα αυτό που κάνουν οι, οι Ρώσοι. Γιατί λοιπόν μπορεί να παραμένει ο φόρο τη ε, κυροζήνη ω μία απειλή γιατί να είναι οι μεταφορές οι σιδηροδρομικές και τόσες άλλες ακριβές ενώ γίνεται όλο και πιο φθηνό το αεροπορικό εισιτήριο γιατί θα πρέπει αυτό να διευκολύνει τις αεροπορικές μεταφορές ε, ώστε να μολύνουν ακόμη περισσότερο. Δεν ε, ισχύουν εδώ κανόνες της αγοράς, απλώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ε, προωθούν αυτή την επιλογή. Αυτές είναι οι συνθήκες πλαισίου, ό,τι και να λέμε. Και πρέπει να το αποδεχθούμε. Και κάτι ακόμη. Ερωτήσεις. Ένας τόνος διοξιδίου του άνθρακα ως εκπομπή. Τι, τι κοστίζει. Τι γίνεται με τα, διοξίδια, με τα οξύδια του αζότου, τι γίνεται με το μεθάνιο, τι γίνεται με, τα άλλα, με τις άλλες χημικές ενώσεις και εκπομπές. Και βεβαίως και μπορούμε να περιορίσουμε τις αεροπορικές μεταφορές, προξενώντας μάλλον δυσκολία σε μια-δυο αεροπορικές εταιρείες, αλλά εν γέννη θα πρέπει οι αεροπορικές μεταφορές στην Ευρώπη να μειωθούν κατά το ίμιση τουλάχιστον για να μειωθεί κατά αξιόλογο λόγο το σύνολο των εκπομπών του δεξιού του άνθρακα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να προσφέρουμε εναλλακτικέ λύσεις μεταφορών για την Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν άλλος δρόμος να διερευνήσουμε, έστω και αν πιστεύω ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό και ρωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πού είναι η εναλλακτική σα. πού είναι η πρώτη εναλλακτική, πού είναι η δεύτερη εναλλακτική, τι γίνεται με τον φόρο προσθέμενη αξία, για τον οποίο δεν είπατε κουβέντα και πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε το φόρο για την κυριοσύνη. Γιατί αυτή είναι η πίεση που ασκείται στην Ευρώπη και περιμένω να δω και οι Ρώσοι, Κινέζοι και Αμερικάνοι πώ θα αντιδράσουν σε αυτά. Φώστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον εισηγητή μας. Τι να πω. Έχω μείνει άφωνη. Εάν τα πράγματα δεν ήταν τόσο ε, ε, σοβαρά, θα το διασκέδαζα κιόλας ακούγοντας αυτά τα χαριτωμένα. Αυτή τη στιγμή η DG ENV ε, κάθετος κλάιμα έρχεται εδώ και μας κουνάει μπροστά από τη μύτη μας κάτι αστείωτητες δεν ξέρω εάν ε, έχει πάθει κάτι όλο το τμήμα και αν ε, έχει πέσει κάποια επιδημία, αλλά σας βεβαιώ ότι είναι γελία αυτά που μας λέτε. Είναι γελιοτάτη η ε, άποψη, η γνωμοδότηση που μόλις μας παρουσιάσατε. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να μετριάσουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και να είμαστε για μία ακόμα φορά εμείς ε, λέει η Κομισιόν θα ξεκινήσουμε στα προφορία, θα έχουμε αποτέλεσμα. Ναι, ενδεχομένως, αλλά ε, δεν ακούτε τι λένε οι άλλες χώρες, γιατί οι άλλες χώρες οι οποίες ε, κυριαρχούν πλέον στον κόσμο ε, τρίβουν τα χέρια τους με μεγάλη χαρά ακούγοντας αυτού του είδους τα μέτρα, γιατί, διαφορετικ... γιατί ούτως ή άλλως εάν τα μέτρα δεν είναι παγκόσμια δεν θα έχουν και καμία επίπτωση. Και εμεί ε, είπαμε να το δούμε και αυτό, να δούμε και αυτή την πτυχή. Ε, και εσεί είπατε εντάξει, να ξανάρθουμε με μια καινούργια πρόταση, αλλά φαίνεται ότι δεν σα αρέσει καθόλου το γεγονό ότι δεν ψηφίσατε, δεν κερδίσατε στην ψηφοφορία. Ε, είχατε ένα 70-30 ε, θέλετε να είσαστε με την ε, πλειοψηφία, αλλά δεν σας άρεσε αυτά που έλεγε η πλειοψηφία, άρα πήγατε από την άλλη πλευρά ε, και τελικά καταλήξαμε σε τούτο εδώ το πράγμα το οποίο είναι απίστευτο. Μιλάμε για ε, αμοιβαία συνένεση. Ναι, αλλά θα πρέπει εδώ να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία δημιουργεί, η οποία προκαλεί στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ούτως ή άλλως μιλάμε για σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς κατηγορηματικά πρέπει να πούμε και το έχουμε πει άλλωστε κύριε Πρόεδρε στο παρελθόν ότι ή θα είναι παγκόσμιο το σύστημα πραγματικά ή διαφορετικά δεν έχει έννοια. Εν πάση περιπτώσει ήδη έχουμε βάλει τους εαυτούς μας σε αυτή τη θέση. Πέραν αυτού τα κράτη-μέλη δεν στηρίζουν αυτά που λέτε. Λέτε τώρα εδώ και ε, ε, κοκορεύεστε, τα κράτη-μέλη συμφωνούν όλα κτλ. Όχι, έχουν βαρεθεί τα κράτη-μέλη με όλη αυτή την κατάσταση, ε, η οποία οδηγεί μαθηματικά σε μείωση της αξιοπιστίας. Μεγάλες χώρες της, του κόσμου ε, ε, λένε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα σωρό καλά πράγματα τα οποία κάνουμε ήδη χωρίς ε, αυτή την γελία νομοθεσία. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτό που σας ενδιαφέρει από ό,τι φαίνεται είναι να έχετε ένα σχεδιάκι, ένα προγραμματάκι και να το προχωρήσετε. Κοιτάξτε, εδώ βλέπουμε κάτι φόρμουλες x, ε, χ ίσον ε, ψ, διά ε, ωμέγα ή οτιδήποτε. Μα αυτού του είδους τις εξισώσεις έχω να τις δω από όταν ήμουν στο σχολείο. Επίσης ακούμε και διάφορες και διάφορες ε, έτσι βαρύγδουπες εκφράσεις του τύπου κύκλος του οποίου η διάμετρος ξεκινάει από το ένα αεροδρόμιο και φτάνει μέχρι το άλλο. Μα τι είναι αυτά τώρα. Τι να σας πω, έχω μείνει άφωνη και νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσετε να παίζετε με τα νεύρα και κυρίως με την ευφυΐα των μελών της Επιτροπής μας. Ε, και πραγματικά, τι να σας πω, δεν καταλαβαίνω τι κάνετε με τις δουλειές που έχετε, δεν καταλαβαίνω με τι ασχολείστε έχοντας τις θέσεις που έχετε. Ε, ε, πραγματικά είναι γελιότητες αυτά που συμβαίνουν και, και τα λέμε εμείς που είμαστε ένας από τους πιο κεντρικούς στο, παίχτες στην παγκόσμια σκηνή. Ελπίζω ότι ο συνάδελφος Κράμερ θα μπορέσει να ε, βγάλει κάτι καλό, να γράψει μια έκθεση η οποία να είναι καλή. Ο, ο Μάικλ προηγουμένως αναφέρθηκε σε plan B, πλαν C, εναλλακτική λύση 1, 2. Ε, ναι, πρέπει να έχουμε τέτοιες εναλλακτικέ και εν πάση περιπτώσει ας, ας δούμε τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος, ας φτάσουμε ε, σε ένα αποτέλεσμα κοινά αποδεκτό, ας φτάσουμε και μέχρι το 2016 εν πάση περιπτώσει, να δούμε τι γίνεται αλλά να προκύψει κάτι το οποίο να είναι σωστό κατά την έννοια του 2020 και να μην αυταπατώμαστε εδώ πέρα. Ε, όταν μιλάμε για τις χώρες, ούτε καν δεν ισχύουν αυτοί οι κανόνες για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν χώρες οι οποίες κατά περίπτωση εξαιρούνται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές ήταν και οι σκέψεις που ήθελα να εκφράσω Μήπως μπορείτε να μου πείτε, εν πάση περιπτώσει, ποιε ακριβώς είναι οι χώρε μέλη οι οποίες στηρίζουν αυτό που κάνετε. Συγκεκριμένα με ονόματα και αριθμούς. Και ε, όπως λέμε και στα αγγλικά, όταν είσαι στο βάθος της τρύπας σταμάτα να, να σκάβεις, μην πας και παρακάτω. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ε, με μεγάλο σεβασμό ακούω όσους έρχονται από την Κομισιόν. Αλλά σιγά σιγά η υπομονή μου μαζί με το σεβασμό μου ε, ε, εξανεμίστηκαν. Γιατί δεν είναι δυνατόν να έρχεται εδώ η Κομισιόν και να μας λέει ψηλολόγια από εδώ, ψηλολόγια από εκεί και να προσπαθείς να οικοδομήσει κάτι. Γιατί μας λέτε ψέματα και σίγουρα δεν μας λέτε σωστά πράγματα. Κοιτάξτε, αυτή η φόρμουλα που μας διάβασες ε, προηγουμένως, τα χύψη δια 100 επί 200 ή ξέρω εγώ τι, ε, βρίσκεται στη, στο τέλος ε, της Κομισιόν μεταξύ Αγγυλών και λέει ότι ε, αυτή η φόρμουλα μάλλον θα διαγραφεί από το τελικό ε, κείμενο ε, και θα αντικατασταθεί από έναν πίνακα αντιστοιχειών που θα έχει εγκριθεί και από την Eurocontrol. Αυτό για να σε παρηγορήσω λίγο, να σε ανακουφίσω λίγο σε αυτό το, το, προβληματισμό που έχεις. Ο κύριος Κόχ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, είναι αυτός σκοπός το ETS, διερωτώ με, ή εξυπηρετεί κάποιον άλλο σκοπό. Διότι ε, εάν θέλουμε να ρυθμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα ε, ελέγχονται οι εκπομπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο μέσα, δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια. Μόνο αν χρειάζεται με τις υπόλοιπες χώρες να ρυθμίσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να ενθαρρύνουμε και τις αεροπορικές εταιρείες να εισαγάγουν πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Αλλά δεν βλέπω αυτό να εξυπηρετείται, ούτε και βλέπω να υπάρχει ένας λόγος να γεμίζουμε τα ταμεία κάποιων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ΙΚΑ τώρα είχε προτείνει σε μία διάσκεψη ένα παγκόσμιο διεθνές σύστημα ε, στηριζόμενο στις αρχές της αγοράς του το 2020. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε όμως λέγοντας «Ε, όσο και να κοστίσει εμείς οπωσδήποτε πρέπει να εισαγάγουμε το σύστημα αυτό. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετούμε τίποτε άλλο από τις αεροπορικές εταιρείε και μάλιστα δεν εξυπηρετούμε καν το στόχο της μείωσης του οξυδιού του άνθρακα. Δεν χρειάζονται λοιπόν ε, τέτοιε λύσει και μάλιστα γραφειοκρατικά βαριές μεταβατικές λύσει. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Και έτσι θα έλεγα stop the clock μέχρι το 2020. Σταματήστε τα ρολόγια. Θέλεις ξανά το λόγο, Μιχαήλ. Εντάξει, θα τον δώσω για λίγο όμως. Μια σύντομη ερώτηση. Θα ήθελα να ξέρω επακριβώς ποια είναι τα νούμερα, το, ο αριθμός μη για τις αεροπορικές μεταφορές στην Ευρώπη. Θέλω ακριβώς αυτά τα στοιχεία να μου τα δώσετε. Okay. Just a few brief questions my... Να κάνω κι εγώ κάποια σύντομα ερωτήματα. Κατά κάποιο τρόπο υποθέτω ότι και εγώ και όσοι ήμασταν εδώ ε, όταν ε, μιλήσαμε για το ETS, νιώσαμε και εμείς κάπως ενοχή για την αμέλειά μας ως μέλη της Επιτροπής Μεταφορών. Είμαι απολύτως πεπισμένος ότι κάναμε λάθος που δεν ζητήσαμε να έχουμε κοινή αρμοδιότητα μαζί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος όταν ε, πρώτο συζητήθηκε αυτό το σύστημα, διότι τότε είχαμε μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Μεταφορών που ουσιαστικά δεν προχώρησε χωρίς τους συναδέλφους από την Επιτροπή Περιβάλλοντος και θα πρέπει οι συνάδελφοι να θυμάστε ότι μπορούμε να ασκούμε κριτική, να ασκούμε κριτική στη Γενική Δεύση για την κλιματική αλλαγή και εγώ ήμουν ο πλέον επικριτικός από όλου σε σχέση με το πώς προχωρεί η κατάσταση. Όμως τελικά υπήρξε συμφωνία στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό μέσω της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Και τα κράτη-μέλη συμφώνησαν. Θα πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη. Από το 2005 ή δεν ξέρω εγώ από πότε και μετά, η πολιτική προτεραιότητα πλέον δεν είναι η διάσωση του πλανήτη, αλλά η διάσωση των θέσεων εργασίας. Σίγουρα ε, ο ε, Μιχαήλ θα είναι απογοητευμένος ε, που τόσο πολύ χαμηλά έχει πέσει ως προτεραιότητα η διάσωση του πλανήτη λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Θα πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι το ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πλειοψηφία το σύστημα αυτό τότε που το ψήφισε. και πριν από τέσσερα χρόνια ε, είχα ήδη μιλήσει για αυτό το εναλλακτικό σχέδιο Plan B δεν υπήρχε κανένα τέτοιο σχέδιο και το ξέραμε. Για ποιο λόγο, διότι τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε αυτό είναι το σχέδιό μας και αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Εμείς όμως από πλευράς μεταφορών δεν αφήνω, ε, αφήνω μάλλον κατά μέρος την Επιτροπή Περιβάλλοντος, εμείς ακούγαμε όλες τις φήμες, τα προβλήματα, τι γινόταν, τι θα γινόταν και εμείς το είχαμε ξεκαθαρίσει και το είχαμε πει τι θα γίνει και έτσι και έγινε. Να το ξαναπώ. Την πατήσαμε. Θα έπρεπε να είχαμε εξασφαλίσει κοινή αρμοδιότητα, κοινή ευθύνη με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και τώρα θερίζουμε ό,τι σπήραμε τότε. Τώρα δεν ξέρω αν ε, έχουμε πέσει στην τρύπα της Τζάκη ή είμαστε στη γωνία κάποιο άλλο. Ε, είπε ο κύριος Κόχ να σταματήσουμε τα ρολόγια και ο κύριος Γκρός θα επιβεβαιώσει ότι σε μια συνεδρίαση που είχαμε πήραμε έτσι κάποια μηνύματα ότι μάλλον δεν θα το δεχθεί το περιβάλλοντος αυτό να σταματήσει το ρολόι. Ε, τι θα πρέπει να κάνει τότε η Κομισιόν, να ψάξει να βρει κάτι άλλο. Και ξέρω ότι αυτό που αναζητεί η Κομισιόν δεν είναι αποδεκτό από όλους. Και υπάρχουν ζητήματα που έχουν προκύψει. Πού πάει όμως η Κομισιόν, ξέρει, εγώ δεν καταλαβαίνω. Και για να τα πω έτσι ντόμπρα και ειλικρινά, όπως λέει και ο Μίχαλ, νομίζω ότι έχει πάρει μια τελείως διαφορετική ε, διαδρομή σε σχέση με αυτό το σύστημα, το σύστημα ε, εμπορίας Αν εμείνει όμως η Κομισιόν σε αυτό το σύστημα, δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Μπορεί τα έρμπα να πηδάνε πάνω και κάτω, να απογειώνονται και να προσγειώνονται όπως ποτέ μέχρι τώρα. Έχουμε και έναν Γάλλο Υπουργό που το ίδιο κάνει, το έχει ξανακάνει, το έχουν ξανακάνει οι Υπουργοί. Η Τζάκη πολύ καλά είπε να μας ε, κατονομάσετε ποια κράτη-μέλη το στηρίζουν αυτό. Εγώ μπορώ να σας πω, Τζάκη, η Γαλλία δεν είναι ικανοποιημένη, αλλά υπάρχει μια εκοφαντική σιωπή αυτή τη στιγμή από τα περισσότερα Τώρα θα μείνει έτσι κατάσταση, θα μείνει έτσι το σύστημα, θα το δούμε. Έχετε λοιπόν εδώ έναν Γερμανό τύπο που έχει ασκήσει έντονες κριτικές ε, στην Κομισιόν για το πώς επεξεργάζεται και για το πώς προχωράμε αυτό το νομοθέτημα το συγκεκριμένο και τώρα επειδή συμπάσχω και συμμερίζομαι τη θέση επιτροπής, εντάξει, εύκολο είναι να το πούμε όλοι αυτό, σας το είχαμε πει, αλλά έτσι δεν θα προχωρήσουμε. Ως Επιτροπή Μεταφορών πρέπει και είμαι σίγουρος ότι και ο Μίχαλη θα κάνει πολύ καλή δουλειά. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα τη συντάξουμε, θα την έχουμε έτοιμη τη γνωμοδότησή μας πριν τα Χριστούγεννα για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε τον Ιανουάριο προτού ψηφίσει η Επιτροπή Περιβάλλοντος. Απλά θεωρώ ότι όλα όσα είπατε ήταν έγκυρα και σωστά, αλλά καλό θα ήταν να θυμόμαστε ποιος τα ψήφισε αυτά στην αρχή. Εμείς τα ψηφίσαμε, τα κράτη-μέλη τα ψήφισαν. Είναι τώρα τα πράγματα σε άθλια κατάσταση, έχουμε σε ένα χάλι περιέλθει, έτσι είναι. Ναι, αλλά τι κάνουμε για να βγούμε από αυτήν την κατάσταση. Ο επικεφαλής του, της, του αεροδρομίου του Μάντσεστερ, ένας καλός μου φίλος, είχε πει ότι όλοι εδώ που είστε γύρω μου μπορείτε να μου πείτε ε, ένα πρόβλημα. Εγώ όμως ψάχνω τον έξυπνο αυτό τύπο που θα μου βρει μια λύση, μια διέξοδο. Και αυτό να ζητούμε κι εμείς. Κυρία Μπάρντραμ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τα σχόλια, για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που ακούστηκαν. Θα προσπαθήσω να ομαδοποιήσω τις απαντήσεις μου. Πρώτα να δούμε την πρόταση που έχουμε μπροστά μας. Δεύτερον, ε, τι προκύπτει από τα σχόλια, δηλαδή ποια είναι η θέση των, τριών, των τρίτων χωρών ε, και τρίτον να κάνουμε μερικές σκέψεις για την συνολική προσέγγιση Global Process. Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι ε, αυτό που προτείνουμε είναι συμβατό με όλες τις συγγενείς οι επηρεαζόμενες πολιτικές, περιβάλλον κτλ. Ε, που έχει καθορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε, ε, είχαμε συναδέλφους, ή μάλλον έχουμε αυτή τη στιγμή στην Βαρσοβία, στις, στη συζητήση για το κλίμα που γίνονται εκεί, συναδέλφους οι οποίοι ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιο είναι το πεδίο ε, στο οποίο, το οποίο μας απασχολεί. Μας απασχολεί βεβαίως και η εξωεταφικότητα ε, και αυτό ε, το μεταφέρουν οι εμπειρογνώμονές μας. Δεν υφίσταται κανείς διακριτική μεταχείριση βάσει της προτάσεως αυτής. Δεν είναι μία πρόταση η οποία έχει γίνει τυχαία. Έχουν γίνει και οι απαραίτητες μελέτες αντικτύπου οι οποίες ε, όντως δείχνουν ότι ε, ε, είναι όντως ελαφρώς επιβαρυντικά τα μέτρα για αυτούς τους αερομεταφορείς που δεν έχουν διευρυμένο δίκτυο μεγάλων αποστάσεων. Πάντως γνωρίζουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί, είναι πραγματοποιήσιμο, είναι βιώσιμο το πρόγραμμα. Κοιτάξτε, οι τρίτες χώρες έχουν ε, υποβάλει ε, γραπτά υπομνήματα ε, στην ΔΟΠΑ υπέρ της προσέγγισης ανά ένα αέριο χώρο αυτή η φόρμουλα την οποία εμείς έχουμε εισαγάγει δίνει την δυνατότητα να βρεθεί ένα σωστός μέσος όρος, μια σωστή αναλογία ε, με τις χώρες οι οποίες είναι στη ΔΟΠΑ αλλά δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι, η άποψη των τριτών χωρών. Κοιτάξτε, οι ε, προτάσεις μας ε, βεβαίως δεν έχουν χαιρετιστεί ιδιαίτερα θετικά, το περιμέναμε αυτό. Η νομοθετική διαδικασία πάντως είναι διαφορετική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το δικαίωμα να νομοθετεί. Οι εταίροι μας ε, στην ε, διεθνή κοινότητα ε, θα πρέπει να, εάν θέλουν να έχουν διεθνείς μεταφορές, διεθνές δίκτυο, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους κανόνες μας που θα βρίσκονται στο δικό μας πλαίσιο. Βεβαίως, με χαρά θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις με τρίτες χώρες όσον αφορά τα τεχνικά ζητήματα, όσον αφορά τους στόχους κτλ. Όμως εμείς θα εφαρμόσουμε το δικό μας, ε, τους δικούς μας κανόνες, τους οποίους θα πρέπει να εφαρμόσουν και οι τρίτες χώρες. Όσον αφορά την Global Process, έχουμε ήδη βρει του, τους πόρους ε, στον προϋπολογισμό για την ανάπτυξη αυτών των παγκόσμιων μέσων. Ε, και στον, στους, ε, στην ομοθεσία μας λέμε ότι θα πρέπει αργότερα να ξανασυζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα συνολικό σχέδιο, global scheme. Επομένως, ε, το patchwork κατά κάποιο τρόπο δεν θα ε, ε, υπονομεύσει το σύστημα. Τώρα, υπάρχουν παρόμοια μέτρα τα οποία ήδη λειτουργούν σε περιφερειακό επίπεδο. Βεβαίως είναι αντιπαραγωγικό να πούμε ότι με την καλή θέληση όλα θα γίνουν και ότι όλα θα γίνουν μέχρι το 2020 τότε, ε, τότε που ε, λαμβάνοντα υπόψη την ε, μεγάλη τάση αύξησης των εκπομπών της αεροπλοείας. Όσον αφορά το stop the clock, Πρέπει να πούμε ότι μιλάμε εδώ για, μια, ε, για ένα σύστημα το οποίο θα λάβει υπόψη το 90% των εκπομπών. Ε, αυτό δεν είναι αμεληταίο και νομίζω ότι όλοι οι εμπορευόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταλαβαίνουν ότι οπουδήποτε ε, εμπορεύονται θα πρέπει να εφαρμόσουν τους κανόνες, τους κατατόπους κανόνες. Uh, plan B. Όσον αφορά την εναλλακτική λύση, κύριε Κράμερ, αυτό το Plan B. Παρατηρήσει εκτό μικροφώνου από τον κύριο Κράμερ, οι διερμηνεί δεν ακούν. Απάντηση τη Κομισιόν. Το πεδίο εφαρμογής ε, θα είναι ε, το 38% αυτή τη στιγμή όμως σε full scope έχουμε 50%. 50% ε, ε, εντός, βρίσκεται εντός του συστήματος εμπορίας ε, εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Επίσης, μεγάλη αύξηση έχουμε και στις ενωσια, ενδοενωσιακές μετακινήσεις. Επίσης θα μπορούσαμε να επιλέξουμε ένα είδος upstream σύστημα εμπορίας ε, εκπομπών με ε, ε, νέα στοιχεία του συστήματος MRB, δηλαδή να μην εφαρμοστεί άμεσα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κοιτάξτε, δεν θα κάνουμε ακρόαση εδώ. Η Είπατε ότι ψήφισε το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη με πλειοψηφία για αυτό το σύστημα ε, εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών. Εμείς όμως σας ρωτήσαμε ε, σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι επικίνδυνη η πρότασή σας για τους κόμβους, γιατί πρέπει βέβαια όπως καταλαβαίνετε να ε, γνωρίζουμε πριν πάρουμε μια απόφαση που θα είναι αρνητική για εμάς. Πρόεδρος. Τζάκι, ε, έθεσες και το ερώτημα τι, λέει, τι λένε τα κρατημέλη, Για τη Γαλλία ξέρουμε, τα άλλα δεν ξέρουμε. Τζάκι, Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, καλή βούληση αν είχατε πάει. Χάθηκε, δεν υπάρχει πλέον. Αυτό είναι το πρώτο και είναι δυστυχές. Ε, δεύτερον, σας είχα, ναι αν μου επιτρέπετε, σας ρώτησα για τις συνέπειες, τις επιπτώσεις. Μπορούμε, ε, ήταν το απορρίψουμε να πούμε ότι κάποιες, ε, κάποιοι κλάδοι με τα που μπορούν να πούν το χ, το ψ και το μέγα. Αλλά δεν αστειευόμαστε εδώ. Ε, έχουμε τις εξαγωγές μας 14 δις δολάρια ε, εμπορεύματα ε, αποκλείστηκαν, είχαν προβλήματα λόγω της Κίνας και τα λοιπά και υπάρχουν και άλλα προβλήματα με ο πρόεδρος. Ακούστε, Πρέπει να επανέλθεις πάνω σε προηγούμενη ερώτησή σου. Ναι, Πρόεδρε, απλά έλεγα ότι δεν υπάρχει ακόμη αναγνώριση των επιπτώσεων των πράξεων της Κομισιόν. Δεν το καταλαβαίνουν, δεν το πιάνουν. Τέλο πάντων, δεν είδα ερώτηση εγώ, λέει ο Πρόεδρος, αλλά ας ακούσουμε τις απαντήσεις στα υπόλοιπα. Για, τις, ε, για τους σταθμούς, τα hub δηλαδή και την ε, ενδεχόμενη αλλαγή πορεία. Το έχουμε υπολογίσει. Θα υπολογίζεται ανάλογα με την ε, απόσταση που διανύεται στον Ευρωπαϊκό ε-, Εναέριο Χώρο. Έχουμε κάνει τη μελέτη επιπτώσεων και διευκρινίζουμε κάποιες λεπτομέρειες ακόμη. Για τις συνέπειες εν στο, στον κλάδο. Ναι, είναι βεβαίως σημαντικά τα μελήματα αυτά, αλλά μην ε, νομίζετε ότι θεωρούμε πως πρόκειται για κάτι το πολύ ε, εύκολο ή το γελίο ή το υποτιμούμε. Το έχουμε πάρει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα υπόψη να έχουμε αξιολογήσει τις απόψεις και των εμπλεκομένων παραγόντων οι οποίες είναι πολύ σημαντικά αποκλίνουσες μεταξύ τους. Αυτή είναι η πρόταση επιτροπής. Είμαστε διαδικασία συν απόφασης και περιμένουμε σχόλια και παρατηρήσεις οι οποίες ασφαλώς θα επηρεαστούν και από άλλους εμπλεκόμενους παράγοντες. Πρόκειται για την ίδια τη φύση της διαδικασίας της συναπόφασης. Και έτσι προχωράμε σε μια επιλογή για την ε, ρύθμιση του κλάδου αυτού σε μια πολιτική η οποία πιστεύουμε ότι θα είναι βιώσιμη και στεναρή. Κοιτάξτε όμως, τρεις φορές σας ρώτησαν οι συνάδελφοι τι γνώμη έχουν τα κράτη-μέλη. Είχαμε μια πρώτη επαφή στο, στην ομάδα εργασίας για το περιβάλλον με τα κράτη-μέλη. Μέχρι τώρα δύο εξ αυτών υπέβαλαν προτάσεις. Άλλα μελετούν ακόμη ποια θα είναι η εθνική τους τοποθέτηση. Νομίζω ότι δίναμε να πω πως τα κράτη-μέλη δείχνουν μεγάλη ευαισθησία στις απόψεις, τοποθετήσεις των τρίτων κρατών. Και εμείς από πλευρά μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για περαιτέρω διαβουλεύσεις με τρίτες χώρες ώστε να ενισχύσουμε την ε, κατανόηση και να ενισχύσουμε και την ίδια την εφαρμογή αυτής της προτάσεως. Πολύ καλή διπλωμάτηση είστε από ό,τι βλέπω από τον Σαμ Τόμκινς στον τελικό του, του κυπέλου. Τέτοιο τάκλινγκ δεν έχω ξαναδεί. Μπράβο σας. Τι να σας πω τώρα, εάν δύο από τα 28 μόνο έχουν απαντήσει, τι να σας πω συγχαρητήρια στα κράτη-μέλη για την επιμέλεια και την, και την δουλειά που κάνουν. Ξέρω ότι δεν θα τολμήσει κανείς εύκολα να σηκώσει το κεφάλι του πάνω από το χαράκομα. αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να μας δώσετε και εμάς κάποιες απαντήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο θα προχωρήσει, θα περάσει διαδικασίε του στο Κοινοβούλιο. Είναι ένα διαφιλονικούμενο ζήτημα και αν φτάσουν Απρίλιο για να αποφασίσουν τα κράτη-μέλη, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι κάθονται με τα χέρια πλεγμένα, πλέκοντας τα δάχτυλά τους και με το στόμα κλειστό και περιμένουν να δουν τι θα πούμε εμείς για να αποφασίσουν αν θα αντιδράσουν. Γι' αυτό λοιπόν κάποιος πια θα πρέπει να βάλει κανένα κεράκι δυναμίτη στα νότα των κρατών μελών, λέει ο ομιλητής, μήπω και κουνηθούν. Φιτιλάκι. Αυτά λοιπόν. Προθεσμίε για τι τροπολογίε, Όχι, για την παρουσίαση του σχεδίου 17 Δεκεμβρίου. Προθεσμία για τροπολογίες θα έχουμε μια-δύο μέρες μετά από αυτό και ψηφοφορία προβλέπουμε για τον Ιανουάριο. Σας ευχαριστώ θερμά ένα κάπως πιο τετριμένο θέμα, Μιχαέλε, ε, συγχώρεσέ μου τον χαρακτηρισμό. Έχουμε να κάνουμε με την παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές. Έχεις το λόγο χωρίς μικρόφωνο. Ε, oh, Ευχαριστώ πολύ, Brian. Νομίζω ότι κολλάει πολύ ωραία στην προηγούμενη συζήτηση γιατί και εκεί, δεν είχαμε, ε, εκεί που δεν είχαμε σημείο B, ε, σχέδιο B, εναλλακτικό σχέδιο και ετηθήκαμε, εδώ μπορεί να έχουμε μεν εναλλακτικό σχέδιο, αλλά επιτυχία δεν έχουμε. Έχουμε ένα θέμα λοιπόν με τι εκπομπέ που δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί. Τουλάχιστον στα αεροπορικέ μεταφορέ το προσπαθήσαμε. Και κάτι, ε, μέχρι τώρα μπορεί να έχουμε καταφέρει τίποτα, αλλά κάτι μπορεί να επιτύχουμε στο μέλλον. Στα ιστελάσει μεταφορέ τίποτα. Εδώ δεν έχουμε φορολόγηση ενεργειακή και προχωράμε χωρίς κανονισμό με 1,47 εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Η συμβολή των πλοίων είναι 30% των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα της ναυτιλίας, πρόκειται για τα πλοία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχουμε περίπου 50.000 θανάτους το χρόνο που αποδίδονται στις εκπομπές του του άνθρακα από την αυτιλία. Δεν κάνουν επαρκές, επαρκείς κινήσεις τα κράτη, οι διεθνείς οργανισμοί για να αντιμετωπίσουν, όπως οι, οι διεθνείς οργάνωση ναυτιλίας, για να αντιμετωπίσουν το μέτρα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και με ακούσει Ματιό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν στη Λευκή Βίβλο. Όχι εσένα, εσένα, γιατί σε επενώ και σε τιμώ με την έκθεσή σου. Προτείνει. Όχι, όχι. Εγώ ίσω τι να πω. 40% λοιπόν μείωση ή δυνατόν έτσι ε, και 50% μέχρι το 2050 για τις εκπομπές. Αυτός ο φιλόδοξος στόχος τον οποίο έχει προτείνει ο εισηγητή μα Ματσιού Γκρό, με μεγάλη πλειοψηφία τον υποστηρίξαμε, δεν έχει βρει ανταπόκριση και αντανάκλαση ούτε καν μέσα στι προτάσει τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η Επιτροπή είναι ακόμα πιο κάτω από αυτή την ε, πρόταση. Και δεν προτείνει σύστημα για διεύρυνση των πιστοποιητικών και για την αυτιλή Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν επιφυλάξει ω προ την διεύρυνση του στήματο ανταλλαγή εκπομπών για την αυτιλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, με όλη αυτή την εμπειρία προτείνει ένα σύστημα για την καταγραφή. Καταγραφή των εκπομπών, όχι για τη μείωσή του. Πριν από 10 χρόνια που ήρθα εγώ στο Κοινοβούλιο, τα ίδια ακούγαμε. Και οι πιο παλιοί, όπω ο Γιαρζεμπόφσκι, μου λέγανε Α, και τα προηγούμενα δέκα χρόνια τα ίδια πάλι λέγαμε. Ε, να λοιπόν. Ε, ακόμα έρχονται για να μα μιλήσουν για καταγραφή εκπομπών, ενώ ξέρουμε τι σημαίνει αυτό ο κίνδυνο των υψηλών εκπομπών του του άνθρακα. Η Επιτροπή λοιπόν δεν επιτελεί το έργο τη, δεν έρεται στο ύψο των υποχρεώσεών τη και μα προτείνει. Μακού, μακού, μακούς» κατά 40% μείωση στο, 50, στο 40% δυνατόν στο 5% για το, μέχρι το 2050 ως εξαιρετική μόνο λύση. Τώρα βλέπουμε ότι οτιδήποτε μπορούμε να κερδίσουμε εδώ στην εσωτερική ρύθμιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύουμε αν δεν επιμείνουμε σχέση με τους εθνείς οργανισμούς να το χάσουμε στη σχέση μας με τις τρίτες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια ε, εξοικονόμηση εκπομπών και πρέπει να σας πω ότι όταν ήταν ακριβά τα καύσιμα, γιατί εκεί παίζεται το παιχνίδι στο κόστος, όταν ήταν ακριβά τα καύσιμα, απλώς πήγαιναν πιο αργά τα πλοία. Κρατούσε το ταξίδι μια, δύο, τρεις μέρες πιο πολύ. Και το ίδιο το έχουμε δει και στα τρένα με μισή ώρα, μια ώρα, δύο ώρες καθυστέρηση δεν επηρεάζεται το κόστος για την εταιρεία, αρκεί να φτάσουν τα εμπορεύματα κάποια στιγμή στο στόχο τους. Έτσι λοιπόν μπορούμε με απλά τέτοια μέτρα, και το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, με μέτρα τα οποία έχουν ήδη σαγάγει για λόγους οικονομικούς και μόνο οι επιχειρήσεις, να εξασφαλίσουμε μέχρι και 75% μείωση των εκπομπών για λόγους ναι, οικονομικού αλλά και οικολογικού εν προκειμένου. Και δεν πρέπει να το μιλήσουμε αυτό. Η μείωση κατά 10% τη ε, ταχύτητα των πλοίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση κατά 19% των εκπομπών. Και σε κόστος λοιπόν, αλλά και σε ε, εκπομπές μπορούμε να κερδίσουμε μόνο από τη μείωση της ταχύτητας. Επίσης αυτό μπορούμε να το συνδυάσουμε με ένα είδος τελών, με ένα οικονομικό κίνητρο, το οποίο θα οδηγήσει τις εταιρείες σε μείωση ταχύτητας, κόστους και, οικολογικής και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. και επαναλαμβάνω ότι μέτρα όπως αυτά των, ε, τα, τα, προτινόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για μερική επιβολή προσθέμενης αξίες, αξίας, ε, αλλά όχι σε όλους, και δεν έχουν καμιά σχέση με την οικονομία της αγοράς, και αποτέλεσμα δεν φέρουν, και δεν μας απαλλάσσουν από τις εκπομπές. Γιατί όταν είναι πιο ακριβό το τρένο θα πάρει κανείς το αεροπλάνο που είναι πιο φθηνό, θα ε, πετάξει και θα μας επιβαρύνει πάλι με το διοξείδιο του άνθρακα και ακόμα χειρότερα. Αν δεν αντιδράσουμε λοιπόν εμείς, αν δεν αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Άρα δεν αντιδράσουν πάνω τα άλλα κράτη στι προτάσει Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κάνουμε. Σε αυτό χρειάζεται μια εναλλακτική λύση. Και παραλαμβάνω, όχι μόνο διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και μικροσωματίδια, Οξίδια του αζότου, μεθάνιο και άλλε λοιπέ ρηπογόνε ουσίε πρέπει να συνυπολογίζονται και να τι περιλάβουμε στο σχέδιο για τον περιορισμό των εκπομπών. Χρειάζεται ένα πλαίσιο χρονικό 2019 είναι μια ημερομηνία πολύ ε, μακριά, θα πρέπει να στραφούμε προς το στόχο του 2016 και πρέπει οι εφοπλιστές, οι οποίοι τους ή ε, από την ε, ε, ναυσιπλοεία ε, ανοιχτής θάλασσας μπορούν να εποφελούνται από ειδικές ρυθμίσεις γιατί βλέπουμε ότι καίνε τα, τα πλοία αυτά στην ανοιχτή θάλασσα, βρώμικο καύσιμο, το πιο ε, δηλητηριώδες, το πιο τοξικό καύσιμο το οποίο εκπέμπουν απλώς όταν βρίσκονται σε ανοιχτή θάλασσα ε, στην ατμόσφαιρα. Ε, αυτοί λοιπόν θα πρέπει να συμβάλλουν με κάποιο τρόπο και ελπίζω ότι θα με υποστηρίξετε στο να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι ε, μεριμνούμε για τα θέματα αυτά και να στείλουμε το μήνυμα αυτό προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκρούς. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου του σκιώδου συζητητού λαμβάνω να μιλήσω. Έχει ξανασυμβεί αυτό αρκετές φορές. Είμαι ο τακτικός θαμών της, πέμπτη, ε, τη συνεδριάσεω τη Πέμπτη. Το ξέρει πια και εσύ, Μπραν. Εδώ μας λέει λοιπόν ο σκιώδης συγητής ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιορίζεται ή θα έπρεπε να περιορίζεται σε περιγραφή των, στόχων και να μην ορίζει εσωτερικούς στόχους. Γιατί προς το παρόν δεν θεωρεί ότι είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Δεύτερον, επισημαίνει και ο ότι όταν στο πλαίσιο των υφισταμένων στόχων, στόχων για ε, φορολόγηση ή για προτίμηση ορισμένων ε, τρόπων μεταφορών. Οι στόχοι ορίζονται, εάν οριστούν μάλλον πολύ υψηλοί, ε, κινδυνεύουμε να περάσουμε και πάλι στις οδικές μεταφορές, να γίνει αυτό το modus shift όπως ονομάζεται, να εγκαταλείψουν την ναυτιλία, ναυσιπλοεία και να περάσουν στις οδικές μεταφορές τα φορτία. Γι' αυτό δεν πρέπει να λησμονούμε αυτήν τη διάσταση και την κατάσταση τη φορολογική, την επιβάρηση φορολογική που ισχύει στα άλλα είδη των μεταφορών. Ιδέτερα δε για τη Βόρεια Ευρώπη και για τις ακτές της είναι πέραν του short, short sea shipping των θαλασσίων μεταφορών μικρών αποστάσεων ε, δυνατή η επιλογή των χερσαίων μεταφορών, κάτι το οποίο βέβαια θα οδηγούσε από τη χέρο όλη την προσπάθεια. Ευχαριστώ. Να πω δύο λόγια ε, πριν δώσω τον, ε, στον κύριο Αρκεντράουι, εδώ μία από μια μια ομαδα του κυρίου Ζαρίμπη από ό,τι φαίνεται εδώ λέει το χαρτί μου ότι είναι senior management αλλά εμένα μου φαίνονται, managers αλλά εμένα μου φαίνονται πολύ νέοι για τόσο για αυτό το βαρύγδουπο τίτλο. Εν πάση περιπτώσει, τους ευχαριστούμε, είναι εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά κρίμα γιατί δεν συζητάμε σήμερα τίποτα για τους σιδηροδρόμους που θα τους ε, απασχολούσε περισσότερο, γιατί είναι από τον τομέα των σιδηροδρόμων. Εν πάση περιπτώσει, σας καλωσορίζουμε και ευχόμαστε να ευχαριστηθείτε εδώ τις συζητήσεις μας. Ο κ. Αλκαντράουι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Θα ήθελα να πω ότι και στη δική μου περίπτωση ο σκιώδης εισηγητής μας ε, απουσιάζει. Θα είμαι λοιπόν πάρα πολύ σύντομος. Ε, νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα, έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ενδελεχέστερα το θέμα αυτό και ε, στο μέλλον. Ο Σκιώδης εισηγητής λέει ότι πρόκειται για ένα πολύ ήπιο ε, βήμα ε, και θα συμφωνήσω και εγώ μαζί του, ε, είναι ένα πρώτο βήμα, εν πάση περιπτώσει, Πάντως ε, είναι ένας καλός στόχος. Εμείς προτιμούμε δεσμευτικούς στόχους και δεσμευτικά όρια όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί γνωρίζετε ότι εδώ η προβληματική προσωμιάζει λίγο με την ε, προβληματική των αεροπορικών μεταφορών. Θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά για να δούμε λίγο πιο μακρόπνοα τι θα ε, κάνουμε στο μέλλον και πέρα από τους στόχους που αφορούν τις ίδιες τις εκπομπές, του σένσου, ε, θα πρέπει να επιμείνουμε να υπάρξουν ε, πρωτοβουλίες ή μέτρα τα οποία θα ε, μειώσουν την ενεργειακή ζήτηση και που επομένως θα μειώσουν και τις εκπομπές. Λυπούμαστε κατά αυτήν την έννοια που δεν υπάρχουν ε, συνολικές προτάσεις, δηλαδή έτσι μια σφαιρική δέσμη η οποία να αναφέρεται σε όλα τα θέματα. Ε, εμείς θα θέλαμε και ε, κάποιες, ε, κάποια μέτρα τα οποία θα αναφέρονται σε διαφορετική χρήση των υλικοτεχνικών υποδομών, διαφορετικά logistics δηλαδή. Βεβαίω δεν θα συμφωνήσουμε με όλες τις λεπτομέρειες που αναφέρονται εδώ, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι σε γενικέ γραμμές συμφωνούμε με το πνεύμα. Ευχαριστώ. Ευτυχώς που δεν κάναμε το λάθος που είχαμε κάνει με την προηγούμενη ε, περίπτωση, δηλαδή δεν έχουμε ε, απολέσει εντελώ κάθε έλεγχο όπως κάνουμε στην περίπτωση του συστήματος ε, πω. Λοιπόν, Κύριε Μάισνερ. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ εκπροσωπώ και ο που απουσιάζει σήμερα. Πριν διαβάσω λοιπόν την τοποθέτησή τη, που την έχει δώσει γραπτό, θα ήθελα να πω ότι ο κύριο Κράμερ, ο οποίο πάντοτε τα έχει καταφέρει πολύ καλά, όπω και σε αυτήν εδώ την γνωμοδότηση, ε, θα πρέπει, επειδή δείχνει μια προτίμηση σε σχέση με την ε, ε, με τι συνδρομικέ μεταφορέ ει βάρο των αεροπορικών, δεν θέλω να του πω ότι όλα τα μεταφορικά, όλα τα είδη των μεταφορών είναι πολύ σημαντικά για μα ιδιαίτερα εδώ στην Επιτροπή των Μεταφορών. Δεν μπορούμε να μειώσουμε, Η να υποβιβάσουμε την αξία της μίας ε, του ενός είδους των μεταφορών εις βάρος μιας του ενό είδου των μεταφορων ει βαρο μια άλλη. Η ισχυώδη συγγήτρια λοιπόν ευχαριστεί τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει και είναι βεβαία ότι θα, κάνουν πολύ, θα είναι πολύ καλή συνεργασία. Ένα δύο σημεία που θα ήθελα να υπογραμμίσω, λέει και ο Δησηγήτρια, είναι τα εξή, ότι συμμερίζομαι με την άποψη ότι δεν είναι η αναμενόμενη σε σχέση με τη Λευκή Βίβλο για τι μεταφορέ η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, οι λύσει, προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2011 που είχαν εγκριθεί μιλούσαν για μείωση των, των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και αντίστοιχα θα πρέπει να ε, δούμε ότι και η οδηγία οδηγεί προς τη μείωση των ε, εκπομπών. Ε, το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι υπερβολικά μακρύ. Γίνεται μόνο πρόταση για επαλήθευση και όχι για μείωση των εκπομπών, όπως την προτείνει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό θα προτιμούσα μαζί με τον εισηγητή να συζητήσουμε μια ουσιαστική λύση. Θέλουμε σαφείς κανόνες για τον κάθε έναν και βέβαια προστασία του θεμητού και υγιούς ανταγωνισμού. θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την προστασία που δεν μας προσέφερε η, οδηγία για το θείο, για το δίκτυο του θείου. Ε, επίσης, ως Επιτροπή των Μεταφορών πρέπει να έχουμε ενημέρωση και πληροφόρηση έγκαιρη και έγκυρη, ώστε να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις, τις καταλληλότερες για τους εμπλεκόμενους, για δε τα είδη των πλοίων που θα καλυφθούν από τον κανονισμό, μπορούμε να συζητήσουμε για τα 5.000 μεικτό μεικτή χωρητικότητα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ικανοποιητική. Τα, τα πλοία αυτά περνούν το περισσότερο χρόνο στα ευρωπαϊκά ύδατα ελιμενιζόμενα ή στα ανοιχτά των λιμένων μας. Και πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Και επίση η πρόταση αυτή θα πρέπει να προωθηθεί σε διεθνέ επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού σε διεθνέ επίπεδο. Αυτά είχε να πει η κυρία Ισηγήτρια. Η κυρία Φώστερ, εκ μέρου του κύριου Βαντάλεν, φαντάζομαι ή μόνοι σας. Όχι, ουσιαστικά θα πω τη δική μου άποψη, γιατί ο κ. δεν είναι εδώ. Συμφωνούμε ότι αυτό το οποίο ζητούμε είναι μια συμφωνία στο πλαίσιο του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού και όχι αυτό μας μα προτείνει εδώ η Κομισιόν. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει πρόβλημα να δει ε, το θέμα της αντιμετώπισης των εκπομπών και άλλα ζητήματα, γιατί σίγουρα θέλουμε να καθαρίσουμε τα αποτέλεσμα των ενεργειών μας. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό είναι κατά ανάγκη ένα σωστός τρόπος να το πράξουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τον εισηγητή, είναι προφανές ότι εργάστηκε πολύ σκληρά. Έχει καταθέσει 63 τροπολογίες. Είμαστε αντίθετοι στις 57. Τις υπόλοιπε 6, έτσι για να σου κάνω ένα δωράκι να σου φτιάξω τη διάθεση, θα τη στηρίξουν. Βελτίωση προς το Μάικλ σε σχέση με το παρελθόν, λέει ο πρόεδρος. Ναι, ναι, πράγματι είναι βελτίωση αλλά για να σοβαρευτώ και λίγο, εκεί που μα δημιουργείται μια ανησυχία και ίσω προέρχεται από την αξιολόγηση των επιπτώσεων, αλλά έχω ακούσει κάποια αριθμητικά στοιχεία από την Κομισιόν και τα βάλε και ο εισηγητή, είναι ότι 50.000 περίπου άνθρωποι πεθαίνουν ω λόγω τη ατμοσφαιρική ρήπανση που οφείλεται σε εκπομπές από τα πλοία. Και πραγματικά ανησυχώ. Όποιο έρχεται εδώ πέρα, στην Επιτροπή μας και μας ε, αναφέρει στοιχεία, χωρίς καμία αιτιολόγηση, και ουσιαστικά το μόνο που θέλουν είναι να υπάρξει ε, μια ανταλλαγή επιχειρημάτων ε, ή καυγάς να προκύψει, δεν είναι αυτό λογικό. Πρέπει να γίνεται μια ανταλλαγή επιχειρημάτων ε, με αιτιολογήσεις. Πράγματι πεθαίνει κόσμος και εγώ που γεννήθηκα στο Λίβερπουλ θα έπρεπε να έχω πεθάνει και εσύ Μπράιον που είμαστε κοντά στη θάλασσα. Άλλο να καθαρίζουμε τη ενέργεια μας και άλλο με αυτόν τον τρόπο. Τέτοια γελία στοιχεία νούμερα τα έχω ακούσει ξανά από την Κομισιό. Να ευχαριστήσω τον Μιχαήλ πάντως για τη σκληρή του δουλειά. Έχουμε μάθει ε, και συμφωνήσει ότι διαφωνούμε σε αυτά τα θέματα. Τέλος πάντων πάμε στο επόμενο στάδιο, Πρόεδρε. I feel... Ευχαριστώ πολύ. Περχόμενος από τη βορειοδυτική Αγγλία, ε, το ότι ζω ακόμα είναι πράγματι ε, κάτι που με χαροποιεί ιδιαίτερα. Η κυρία Μπάλτρομ από την Κομισιόν. Uh, and, uh, indeed. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τα σχόλιά τους. Έχουμε μελετήσει με ενδιαφέρον ε, την έκθεση του εισηγητή σας. Σε μια πρώτη φάση τι περιμένουμε και αυτή τη απογοήτες που εκφράσατε. Αυτό το σχέδιο ΠΙΕ e, δηλαδή παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων και εξακριβώς θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα προς μια πιο συνολική προσέγγιση. Πριν από κάποια χρόνια ε, είχαμε πει ότι θα πρέπει ο ναυτιλιακός τομέας να συμπεριληφθεί στο σύστημα ανταλλαγής δικαιωμάτων εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκτοτε υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, που είναι ένας κεντρικός οργανισμός για να προωθήσει αυτό το θεματολόγιο και ιδίω σε ό,τι αφορά το MRV, αυτό το σύστημα παρακολούθησης υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης, που ξεκίνησε πολύ καλά με βάση την Αμερικανική πρόταση που την επεξεργάζονται οι ομάδες των εμπειρογνωμόνων περαιτέρω αυτή τη στιγμή. Εμεί Εμείς θέλουμε να συμβάλλουμε θετικά στις ε, διεθνείς αυτές, αυτές συνομιλίες, χωρίς να προεξοφλήσουμε ε, την πρόοδο που θα πρέπει να επιτευχθεί σε διεθνές επίπεδο περιμένουμε να έχουμε σημαντικούς σταθμούς, ορόσημα από πλευράς ναυλιακών από τα επόμενα χρόνια. Και θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε το χρονοδιάγραμμά μας και εμείς, ότι αφορά των προτάσεών μας. Βλέπουμε ότι τα επόμενα βήματα που προβλέπονται, παραδείγματος χάρη ένα σύστημα force charging system, θα απαιτήσει νέα πρωτοβουλία από την Κομισιόν και μια αξιολόγηση επιπτώσεως. Ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή, από τεχνικής πλευράς δεν είναι εφικτό εμείς να προχωρήσουμε στις διαπιστεύσεις των επαληθευτών ε, για το MRV πιο γρήγορα. Κάνουμε ότι είναι και πρακτικά και τεχνικά εφικτό. Σε ό,τι αφορά την ε, διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής για να καλυφθούν και άλλοι ρήποι. Καταρχήν συμφωνούμε ότι η παρακολούθηση των ρήπων είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν υπάρχει όμως μηχανισμός ή μέθοδος αυτή τη στιγμή για να ελέγχουμε αυτούς τους ρήπους. Δεν νομίζουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να καθυστερήσει η παρακολούθηση των εκπομπών διεξουδίου του άνθρακα βάση αυτών. Είδα όμως σε αιτωικές ε, σκέψεις ότι ε, υπάρχει αυτή η διάθεση, ένα άνοιγμα δηλαδή για να ληφθούν υπόψη και άλλοι ρήποι στο πλαίσιο μιας παρόμοιας προσέγγισης εφόσον υπάρξουν τεχνολογίες σχετικές και εξοπλισμός ανάλογος. Θα μπορούσαμε να τα εντάξουμε δηλαδή, να εντάξουμε αυτούς τους ρήπους. Προσεχώς, ό,τι αφορά τώρα ε, τα κατόφλια ε, για τα, τις τιμές, δηλαδή τις ωραίες τιμές, ποια πλοία θα καλύπτονται, αυτά γίνονται ε, στο πλαίσιο του ε, IMO, 400 γιγατόνι συζήτηση στο πλαίσιο του Διεθνούς Αθλητικού Οργανισμού. Θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση, αλλά λαμβάνοντα υπόψη ότι θα πρέπει και διοικητικά, διαχειριστικά να είναι ανάλογο αυτό το οποίο θα προτείνουμε. Η αύξηση, η μείωση ε, της τιμή τιμής θα αυξήσει τον, ε, το ποσοστό ε, των πλοίων του στόλου που καλύπτονται από 55 σε πάνω από 90 αλλά δεν θα είναι και αντίστοιχα μεγάλο το ποσοστό ε, του διοξιδίου του άνθρακα που θα καλυφθεί, γύρω στο 5% παραπάνω. Αυτά πρέπει να τα έχουμε όλα υπόψη μας. Με αυτά τα σχόλια νομίζω ότι θα σταματήσω. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Μίχαελ, κάποια αντίδραση. Ναι και ευχαριστώ βεβαίω για τις τοποθετήσεις και για την μεγάλη υποστήριξη που δεν περίμενα. Συμφωνούμε απολύτως, αγαπητή κυρία Μάισνερ. Δεν θέλω μόνο σιδηρόδρομο. Το 80% των, ε, θαλασσι... Ε, πλωτών μεταφορών περνάνε από το Ρήνο στην Ευρώπη. Αλλά δεν θέλω και ε, τα χρήματα να πηγαίνουν μόνο σε ένα μέρος. Όταν προσαρμοστούν τα πλοία λοιπόν στις ανάγκες και τις συνθήκες των πλωτών μεταφορών μέσα από ποτάμια και αντίστοιχα πάνε και τα, τα λεφτά εκεί που πρέπει για να υποστηρίξουν αυτές τις μεταφορές, ναι. Αλλά αυτό που γίνεται είναι ότι ε, δεν έχουν δοθεί λύσεις για πολλούς τύπους ε, εκπομπών που υπάρχει δυνατότητα να μετρηθούν. Τεχνολογικά η επιστήμη το προσφέρει αυτό, το επιτρέπει. Η Επιτροπή μας είπε ότι μίλησε με κάποιους κατασκευαστές. Ε, γιατί δεν έχουμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Και γι' αυτό χαίρομαι που η συνάδελφό σου υποστηρίζει αυτές τις προτάσεις ξέρει πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση με την βόρεια θάλασσα και τις ε, θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για τη βόρεια θάλασσα και σε άλλες περιοχές θα πρέπει αντίστοιχα να μελετήσουμε προσεκτικά την κατάσταση και ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και εσένα και την ομάδα σου. Surprise! Υπέροχη έκπληξη κυρία Φώστερ που με υποστηρίζετε κι εσείς. Και τελευταία παρατήρηση και αυτό μια μορφή τακτικής επιλογής είναι, ξέρετε. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολείπεται τόσο πολύ των επιλογών των δικών μας, τότε θα μπορούσατε να πείτε σε σχέση με το Συμβούλιο, μα αυτοί, ε, αυτοί συμφωνήσανε και εμείς ε, δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Αλλά εδώ πέρα μπορείτε ωραιότατα να προχωρήσετε ακόμη περισσότερο. Έχετε και την ε, τεχνογνωσία, έχετε και τα μέσα, πολιτική και τακτικές επιλογές έστω. Εάν όμως εκ προημίου έχουμε τόσο χαμηλά ορίσει τον πύχη, δεν μπορούμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα. Γι' αυτό θέλω να πω να είστε πιο φιλόδοξοι, more ambitious και να προσφέρετε λύσεις οι οποίες είναι πιο κοντά σε αυτά που έχει επιλέξει το Κοινοβούλιο για να προχωρήσουμε και πιο καλά. Ιδάλλως ούτε το Συμβούλιο θα προχωρήσει πιο πέρα. Αυτά και περιμένω με χαρά τις τη συζητήσεις. Ευχαριστώ, Λεπρόεδρος. Η προθεσμία για τις τροπολογίες υπενθυμίζω 3 Δεκεμβρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 21 Ιανουαρίου. Τροπολογίες 3 Δεκεμβρίου. Ψηφοφορία στην ΤΡΑΝΑ 21 Ιανουαρίου. Στο επόμενο θέμα. Ενιαία Ευρωπαϊκή Ουρανή. Αναδιατύπωση. Κύριε Γκρός εκ μέρους του κυρίου Μαρινέσκου και μετά θα ακούσουμε τον κύριο Σασόλη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαρινέσκου δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι παρόν. Έχει ετοιμάσει ένα σύντομο ε, υπόμνημα. Ευτυχώ όχι στα ρουμάνικα, γιατί θα είχα κάποια δυσκολία να σας το διαβάσω στα γαλλικά. Και μας λέει λοιπόν στα γαλλικά ότι εδώ. Και πέντε χρόνια τίποτα θεαματικό δεν έχει γίνει και ε, ε, προς έκπληξή μας ε, στην ουσία το δεύτερο πρόγραμμα έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στα κράτη-μέλη, ε, διότι δεν επιτρέπει μια ε, καλή και συνολική προσέγγιση του τομέα. Ε, πρέπει να πούμε ότι και η πρόθεση που έχει κάνει το Συμβούλιο μέχρι τώρα είναι μάλλον διοικητική φύσεως. Ο εισηγητής προτείνει μια άλλη προσέγγιση, δηλαδή μια προσέγγιση top-down και όχι αυτήν που είχαμε μέχρι τώρα, δηλαδή την από κάτω προς τα πάνω τα κύρια σημεία της έκθεσης του είναι από τη μία πλευρά η ανεξαρτησία των εποπτικών αρχών. Εδώ θεωρεί λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει μονάχα μία ε, ε, αρχή, μία ενιαία αρχή όσον αφορά το Future Air Block θεωρεί ότι θα πρέπει να αφήσουμε αυτή την επιλογή γιατί μόνο χρήματα μας κοστίζει. Όσον αφορά το unbundling ε, ε, θα πρέπει το degroupage λέγεται στα γαλλικά ε, θεωρεί ότι ε, δεν θα πρέπει να προωθηθεί κυρίως η θεωρία αλλά περισσότερο η πράξη ε, και η συνεργασία, η αγαστή μεταξύ των δύο ε, σκελών να, είναι, να προωθηθεί πραγματικά οι στόχοι έτσι όπως έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή θα πρέπει να ε, οδηγούνται και από κοινή συζήτηση με ε, τα κράτη-μέλη. Επίσης ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να προωθεί και τεχνική ΣΕΖΑ Επίσης θα πρέπει να αποσαφινιστεί ε, το πρόγραμμα ΣΕΖΑ, θα πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι ε, οι ε, χρήστες και πώς θα ελέγχονται. Θα ήθελα εγώ προσωπικό τώρα να συμπληρώσω ορισμένα λόγια για τα όσα λέει ο κύριος Μαρινέσκου ότι αντίθετα από τον συνάδελφο θεωρώ ότι δεν ήταν η χειρότερη λύση η αλλά ότι αντιμετώπισε την κακή διάθεση των κρατών και γι' αυτό δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Εάν θέλουμε λοιπόν να εξαρχίσει να δούμε το θέμα, νομίζω ότι οφείλουμε και μπορούμε να επανέλθουμε στους στόχους που είχαμε καταγράψει με το σύστημα ανταλλαγών και άρα μπορούμε να ζητήσουμε μια σαφή εφαρμογή της απόφασης. Και να κοιτάξουμε να επιδιώξουμε πρόοδο που θα ξεπερνάει την απλή οικονομική, το απλό οικονομικό κέρδος από το σύστημα της ανταλλαγή. Σε αυτό νομίζω θα πρέπει να βοηθήσουν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να επιδείξουμε μια σαφή βούληση συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί και οικονομικά είναι συμφέρον και ε, πιο ασφαλές το κρίνο και βέβαια οικολογικά πιο ε, καθαρό. Ανεξαρτήτως λοιπόν των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις οποίες εγώ κρίνω πολύ μετριοπαθείς, πρέπει νομίζω να αναφερθούμε στην εφαρμογή του συστήματος που υπήρχε ήδη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή που καλύπτει το τμήμα ΕΑΣΑ, ε, ΕΟΑ δηλαδή, ο κύριος Ασόλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο κανονισμός για τα αεροδρόμια, τη διαχείριση της ενέργειας κυκλοφορίας και της υπηρεσίας αεροναυτιλίας αποτελεί, όπως γνωρίζετε, μέρος της δέσμης για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και αντιμετωπίζει το ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την εναέρια ασφάλεια, καθώς επίσης και με τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Αεροπορίας, της ΕΑΣΑ δηλαδή. Πρόκειται στην ουσία για έναν κανονισμό το που είναι πολύ τεχνικός, αλλά οπωσδήποτε αντιμετωπίζει και το κεντρικό ε, θέμα της διακυβέρνησης ε, του οργανισμού. Το κείμενο ε, μπορεί να χωριστεί σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά ε, την, ε, τον, ε, την προσαρμογή στον ενιαίο ουρανό, την ασφάλεια και την διαχείριση. Το δεύτερο τμήμα αφορά την αναθεώρηση της διακυβέρνησης του οργανισμού ε, βάση της Διοργανικής ε, Συμφωνίας ε, για τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς του Ιουλίου 2012. Ε, προσωπικά θεώρησα ότι δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθώ με το τεχνικό μέρος του κανονισμού, έχοντας μάλιστα ακούσει και διάφορου, διάφορες παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους εμπλεκόμενους ενδιαφερόμενους ε, φορείς. Θεώρησα ότι η συνένεση είναι καθολική επί του κειμένου της ε, Κομισιόν. Ε, μάλιστα με προσθήκη πέραν των προβλεπωμένων του κανονισμού 216-2008 ε, και υπηρεσιών ATM, δηλαδή διαχείριση εναέρειας κυκλοφορίας, καθώς επίσης και υπηρεσίες ANS, ε, δηλαδή αεροναυτικές πληροφορίες, πλοήγησης, εποπτείας κτλ. Θα ήθελα να ασχοληθώ με τη διακυβέρνηση του οργανισμού. Η Κομισιόν έχει υποβάλει μία μάλλον καινοτόμα ε, πρόταση διότι προβλέπει την αναθεώρηση του ίδιου του οργανισμού βάσει της αναδιανομής ε, των ε, αρμοδιοτήτων που θα βασίζεται στην εποπτεία των, ε, της ασφάλειας ε, καθώς επίσης ε, και του τεχνικού μέρους και από την άλλη πλευρά θα υπάρχει βεβαίως και η Ευρωκοντρόλ που που θα ασχοληθεί με τα επιχειρησιακά καθήκοντα. Ε, έγινε και μια πρόταση τροποποίησης του τίτλου ε, έτσι ώστε να δοθεί η εντύπωση ότι ε, ο οργανισμός παίζει κεντρικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην ουσία όμως βγάζοντας τη λέξη ασφάλεια ε, τροποποιεί κατά κάποιο τρόπο τον ρόλο του οργανισμού. Εγώ θα συμφωνήσω με την άποψη της Κομισιόν για τον νέο ρόλο του οργανισμού γιατί θεωρώ, ότι είναι ένα πρώτο βήμα έτσι ώστε να γίνει κύριος πρωταγωνιστής σε ένα όλο και μεταβαλλόμενο και όλο πιο ε, απαιτητικό παγκόσμιο ε, σύστημα και επομένως αλλάζουν οι αρμοδιότητες, αλλάζει και το όνομα. Πρότεινα λοιπόν πρόταση αλλαγής ε, στο ε, κείμενο της Κομισιόν ε, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να ξαναμπεί η λέξη ασφάλεια. Τούτη τη στιγμή υπάρχουν και διμερείς σχέσεις με, άλλους σημαντικ... με άλλες σημαντικές χώρες όπως είναι ο Καναδάς, η Σιγκαπούρη, το Ισραήλ στον τομέα τη αεροπλοεία πάντα και επομένως ε, δεν θέλουμε μονάχα την απλή ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά την ε, μαύρη λίστα, την black list των παγκόσμιων ε, εταιριών, αλλά θέλουμε και ανταλλαγή βελτίστων πρακτικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη ακόμα ασφάλεια της αεροπλοείας και μεγαλύτερη διασύνδεση των εμπλεκομένων φορέων της Διεθνούς Όσον αφορά την διακυβέρνηση, η Κομισιόν θέλησε να υλοποιήσει την νέα διοργανική συμφωνία του Ιουλίου 2012, όπως είπα και προηγουμένως. Σύμφωνα με, την, ε, με τη συμφωνία αυτή, η Κομισιόν, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν επιτύχει συμφωνία επί της κοινής προσέγγισης για, ε, για τους Πρόκειται για συμφωνία η οποία ε, ενώ δεν είναι ε, δεσμευτική ε, ε, και βασίζεται σε προσέγγιση αναπερίπτωση, παρόλα αυτά λαμβάνει υπόψη πολλά στοιχεία. Τη δημιουργία των οργανισμών, την επιλογή της έδρας, την διακυβέρνηση την λειτουργία τους, την χρήση ε, των πόρων, καθώς επίσης ε, και τον τρόπο με τον οποίο ε, λαμβάνει η χώρα ο έλεγχος. Πρόκειται για στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία αφορούν με σημαντικούς οργανισμούς που εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι σημαντικό να συμμετέχει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή και επομένως φρονούμε ότι είναι σημαντικό ο ε, διοικητής του οργανισμού ε, να λογοδοτεί ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, είναι εξίσου σημαντικό το Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, όπου εκπροσωπούνται τα διάφορα κράτη-μέλη, είναι σημαντικό, λέω, ε, να υπάρχει μία ανακύκληση η οποία ε, θα δίνει την δυνατότητα σημαντικής εκπροσώπησης αλλά ε, και χρονική εναλλαγή η οποία θα επιτρέπει ταυτόχρονα και την επιχειρησιακή συνέχεια. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει να μας, να, ε, ε, μας απασχολήσει είναι οι νέες αρμοδιότητες οι οποίες θα περάσουν από το Ευρωκοντρόλ στον οργανισμό. Αυτό είναι ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, διότι η αύξηση του προϋπολογισμού του οργανισμού θα σήμαινε δημιουργία προηγουμένου ε, και είναι μηχανισμός επικίνδυνος διότι και άλλοι οργανισμοί θα μπορούσαν αντιστοίχως να ζητήσουν αύξηση του προϋπολογισμού. Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί μέσω μεταθέσεως της γραμμής του προϋπολογισμού ε, και ταυτόχρονης επομένως ε, μετάθεσης των πόρων τα οποία χρησιμοποιούνται πριν ε, για, για την πληρωμή των υπηρεσιών ATM, δηλαδή υπηρεσίες νέας κυκλοφορίας, στο τη μετατοπίσή τους λέω στο Eurocontrol. Τέλος, τελευταίο σημείο, είναι αυτό το οποίο αφορά τις εκτελεστικές πράξεις και τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Υπενθυμίζω ότι ε, σχετίζονται μονάχα με τα τεχνικά ε, χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει τακτικά να επικαιροποιούνται και να συμπληρώνονται έτσι ώστε να ακολουθηθούν οι διεθνείς τεχνικές πρακτικές. Βεβαίως παραμένω στη διάθεσή σας έτσι ώστε ε, να λάβω υπόψη μου τις ε, προτάσεις τροπολογίας ε, τις οποίες ενδεχομένως έχετε να υποβάλλετε. Θα έχω σύντομα και συνάντηση με τους σκιώδεις εισηγητές έτσι ώστε να συζητήσουμε θέματα τα οποία σχετίζονται και με τη διακυβέρνηση και με τις τεχνικές, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οργάνωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ε, ούτως ή άλλω οι σκιώδει είναι ίδιοι και για τις ε, δύο εκθέσεις. Ε, Μάικλ, θέλει ε, να ξαναπάρει το λόγο. Ο κύριο Δανέλη, λοιπόν, να ξεκινήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ολοκλήρωση του ενιαίου αφορά στην ποιότητα και στο κόστο των αερομεταφορών που απολαμβάνουν οι πολίτε. Αφορά στην ανταγωνιστικότητα και άρα τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού τομέα αερομεταφορών. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι διατηρούμε ακόμα 28 διαφορετικά συστήματα τα οποία είναι και ασύμβατα μεταξύ τους αεροναυτιλίας και 60 διαφορετικά κέντρα ελέγχου. Ε, πρόκειται για μια προφανώς απαράδεκτη κατάσταση. Γι' αυτό άλλωστε στο Κοινοβούλιο υπάρχει ευρύτατη συνένεση όσον αφορά τη χρησιμότητα του νέου πακέτου μέτρων. Σε γενικές γραμμές η κατεύθυνση της Κομισιόν όπως και του εισηγητή είναι σωστές ε, θα θέλαμε όμως, αποδεχόμενοι ότι βελτιώνουν και επιχειροποιούν ένα πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο, να ε, αναφερθούμε σε κάποιες διαφορές μας. Η Επιτροπή προσπάθησε με την πρότασή της για το διαχωρισμό των υποστηρικτικών υπηρεσιών να εξαναγκάσει τους παρόχους να προχωρήσουν σε μια μαζική και ταυτόχρονη απελευθέρωση. Αυτή η πρόταση δεν ήταν ρεαλιστική και γι' αυτό συμφωνούμε με τον εισηγητή που αποσύρει την πρόταση αυτή στην έκθεσή του. Η απελευθέρωση των υπηρεσιών αυτών δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αυτός Ο διαχωρισμός που προτείνεται θα ήταν περίπλοκος και θα απαιτούσε νέες διαδικασίες με απρόβλεπτο αντίκτυπο και στη λειτουργία αλλά και στο κόστος του συστήματος. Εδώ λοιπόν πρέπει να εξετάσουμε κάποιες αναλλακτικέ προσεγγίσεις. Επιπλέον, προτάσεις του εισηγητή που χρειάζονται αποσαφήνιση περιλαμβάνουν το ρόλο της ΕΑΣΑ, τις εθνικές αρχές και το άρθρο 9 για τις αναθέσεις. Για τα τεχνολογικά ζητήματα και συγκεκριμένα τις τροπολογίες 95 και 97 θα ήταν προτιμότερο να μπουν στον επερχόμενο κανονισμό για το ΣΕΖΑΡ και πιθανώς όχι εδώ. Όσον αφορά τις εθνικές αρχές, οι προτάσεις της Επιτροπής και του εισηγητή κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα προσπαθήσουμε να συνθέσουμε κάποια ακόμη ισχυρότερα μέτρα για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους. Θα θέλαμε να δούμε επίσης μεγαλύτερη διαφάνεια στους παρόχους υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Τέλος, πρέπει ο ανθρώπινος παράγοντας να βρει έκφραση μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο, για παράδειγμα στο μηχανισμό επιδόσεων. Κριτήρια που αφορούν το προσωπικό μπορούν να εφαρμοστούν με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας, αλλά και την ομαλή προσαρμογή στις τεχνολογίες του ΣΕΖΑΡ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους εισηγητές και τον κύριο Μαρουνέσκο Ερήμην βεβαίως. Στους ε, ευρωπαϊκούς ουρανούς είμαστε πια πολύ ανυπόμονοι. Γιατί έπρεπε να έχει οριστεί ημερομηνία εδώ και καιρό. Και βλέπουμε ότι τίποτε δεν έχει γίνει, τουλάχιστον επισήμως. Γι' αυτό αντιλαμβάνομαι ότι έχει κάνει μια επιπλέον πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και πάλι θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ε, τα στοιχεία πέρσι του Δεκεμβρίου που είχαν ε, συμφωνηθεί ότι έχουμε προχωρήσει σε σχέση με το ΦΑΠΣ, ότι έχουν ε, υπάρξει κάποιες ενδείξεις συμφωνίας. Τώρα, ωστόσο, αυτά δεν αρκούν. Χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στους ευρωπαϊκούς ουρανούς και όπως είπε και ο κύριος Σασόλη, Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε πλέον αυτή τη στιγμή να ανεχθούμε. Τώρα, το τι ρόλο θα διαδραματίσει η Eurocontrol, η IAT και όλοι αυτοί θα δούμε. με το FAPS μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Δεν εμποδίζει τίποτε δηλαδή αυτούς, τον προσδορισμό αυτών των ρόλων. Και επίση μπορούμε να δούμε χώρε όπω η, Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία πώ μπορούν ενδεχομένω να δραματίσουν ένα πρωτοποριακό ρόλο για να προωθήσουν τη λύση. Επίση, σε όσα είπε ο κύριο Μαρινέσκου με την έκφραση διάσκεψη των υπουργών στο Βίλνιους, το Φαπ τέλειωσε, έληξε, χρειάζεται νέα λύση. Δεν ξέρω πρέπει να είμαστε τόσο ριζοσπαστικοί, τόσο ακραίοι. Δεν θα πρέπει μήπως να διεκδικήσουμε μια λύση ως το δυνατόν πιο γρήγορα. Και συζητώντας με τον κύριο Μαρινέσκου θα προσπαθήσω να δω μαζί του εάν το top-down είναι η καλύτερη λύση, εάν μπορούμε από τη βάση ξεκινώντας να βρούμε μια λύση. Αλλά το βασικό πάνω απ' όλα να βρούμε μια λύση που θα φέρει αποτελέσματα, που θα λειτουργεί. πάντα μιλούμε για αποτελεσματικότητα. Και τελικά αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να λέμε ότι τα μεγάλα κράτη πρέπει να κάνουν τη μεγάλη προσπάθεια και τα μικρότερα απλώ να βολευτούν. Ε, Όμω αυτό δεν νομίζω ότι αρκεί. Θα πρέπει να βρούμε μια λύση λογική η οποία θα ορίζει βεβαίω την ευθύνη για το κάθε κράτο μέλο και το μερίδιο τη ευθύνη, αλλά που θα έχει και μια πιο ισότιμη κατανομή και αναλόγω θα δούμε τι είδου θεσμικά τι είδους λύσεις μπορούμε να δώσουμε, πώς μπορούμε να εξυγχρονίσουμε, πώς μπορούμε να επικαιροποιήσουμε όλη αυτή τη ε, λύση. Αυτά με τις δύο εκθέσεις που αποτελούν πιστεύω μια πολύ καλή βάση για πρόταση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ Κράμερ. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας Λίχτενμπεργκερ, της κοιόδους συγγήτριάς μας. Εχθές ε, ήταν στην ε, Γερμανία για να συζητήσει το θέμα των διοδίων για τους αλλοδαπούς. Ξέρετε, δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα έρθει να συζητήσουμε κάτι τέτοιο στη Γερμανία, αλλά ήρθε φέρεται η στιγμή ακόμη και γι' αυτό. Για τον κύριο Γκρός. Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί του. Έχουμε να κάνουμε μια win-win-win situation και σε, τρία επίπεδα κερδίζουμε και εξοικονομούμε κόστος και περιορίζουμε τις εκπομπές και ενισχύουμε την ασφάλεια. Και εφόσον λοιπόν η Ευρώπη δεν, εάν η Ευρώπη δεν μπορέσει να επιφέρει αυτή την, ε, το τριπλό κέρδος, αυτή την τριπλή θετική λύση, τότε τι να την κάνουμε και την Ευρώπη και την Επιτροπή. Δεν χρειάζονται. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση με τόσο ακραία θετική πρόταση να μην προχωρήσει. Και ήδη από πέρσι τα κράτη τα οποία έχουν τοποθετηθεί και εδώ δεν μιλάμε πλέον για περιεχόμενο. Μιλάμε για το που έχουν υπογράψει τα κράτη, δεν μιλάμε πλέον για περιεχόμενο, για ουσία. Μιλάμε για το αν η Ευρώπη είναι ένα κράτο δικαίου. Είναι ένα χώρο δικαίου και αν ισχύει ο νόμο. Έχετε υπογράψει, έχετε συμφωνήσει, έχετε δεχθεί όλε αυτέ τι συμφωνίε και συμβάσει και τώρα τα αγνοείτε όλα αυτά. Δεν πειράζει και η υπογραφή που βάλαμε. Τα αγνοούμε όλα. Ξαναρχίζουμε από την αρχή τη συζήτηση. Αυτό είναι τεράστιο κίνδυνο για ολόκληρο το εγχείρημα που ονομάζεται Ευρώπη. Εάν περάσει αυτή η τοποθέτηση ένας συντονιστής που είναι γνωστός σε όλους μας, ο Γεώργια Αζεμπόφσκι, ο οποίος βεβαίως με όλες τις διαφορές μας στην ε, ε, πολιτική των μεταφορών έχει τοποθετηθεί και, έχει, και ήταν ο καταλληλότερος διαπραγματευτής εκ μέρους του Κοινοβουλίου, δεν μπορεί κανείς να τον αμφισβητήσει αυτό. Ναι, κυρία Μάιστερ λέει, ευχαριστούμε. Ναι, βεβαίω και τον υποστήριξα. Βεβαίω και προωθώ αυτέ τι θέσει. Ήταν και νομικό εξάλλου. Ήταν δεδομένο ότι θα είχε τι καλύτερε προτάσει. Δεν, δεν χωρί συζήτηση. Και τώρα να μα λέει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υπάρχουν πια αυτέ οι συμφωνίε, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί όλα αυτά. Εδώ είναι η ώρα να δούμε τι έχει να πει ο καθένας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει ό,τι προτάσεις θέλει, αλλά πρέπει πάνω απ' όλα να μεριμνά για την τήρηση των νόμων, των συμφωνιών, των υπογραφών. Εάν δεν το πράξει αυτό ο θεματοφύλακα, δεν καταλαβαίνω τι ρόλο εξυπηρετεί η έννοια του κράτου δικαίου. Βεβαίω είναι πολύ σημαντικά τα συστήματα που μας προτείνεται ε, να μην υπάρχουν ε, προβλήματα ως προς την ε, ε, συμφόρηση των μεταφορών, αυτό το έχουμε δει και ε, με τους σιδηροδρόμους, μπορούμε να το κάνουμε και με τις αεροπορικές μεταφορές, πρέπει να κοιτάξουμε τις εκπομπές βεβαίως, αλλά μπορούμε και κονδύλια και ε, να εξοικονομήσουμε και από τη ρήπανση να δούμε σημαντική μείωση και να βελτιώσουμε την ασφάλεια. Αφού υπάρχουν αυτές οι συμφωνίες λοιπόν πρέπει να επιμείνουμε, πρέπει να εφαρμοστούν πάκτα sunt σερβάντα. Το είχε πει και ο Φραντς Ιώζεφ Στράους, ο ίδιος εκείνος ο Φραντς Ιώζεφ Στράους, ο οποίος παραβίαζε τακτικά όποια συμφωνία είχε συνάψει, αλλά εν περιπτώσει αυτό ισχύει από αρχαιοτά των χρόνων. Πάκτα σουν σερβάντα. Κύριε ευχαριστώ κύριε Φώστερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα συμφωνήσω σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Μίχαηλ. Θυμάστε ότι ξεκίνησε με δική μου έκθεση της πρωτοβουλίας για τον Γκέοργ Γιαζεμπόφσκι Μήπω τον παρέτησαν, γιατί εξαφανίστηκε. Παντώ ήταν πράγματι ένα πολύ καλό σύμμαχο σε όλη αυτή τη δουλειά για τα ΦΑΠΣ. σω θα μπορούσε να μα ενημερώσει η Επιτροπή, να μα πει τι συνέβη στον καλό μα συνάδελφο τον Γκέορκ διότι συμφωνώ, χωρί ε, να θέλω να σα παγορεύσω τίποτα, αλλά με την ιδιότητά μου ω ε, Βρετανίδας, ε, εμείς για το ΣΕΖΑΡ και για τον Ενιό, για Ευρωπαϊκό είμαστε από του καπανεί και το προωθούμε και το πιέζουμε το θέμα εδώ και καιρό. Έχουμε βέβαια το πράσινο θεματολόγιο, αυτά τα ζητήματα ανταγωνισμού και όλα αυτά, αλλά σίγουρα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση στον ε, χώρο αυτό, τον ενέριο που έχει μεγάλη, παρουσιάζει μεγάλη συμφόρηση. Ό,τι αφορά την έκθεση Μαρινέσκου πράγματι, ε, πολύ μεγάλο μέρος της είναι καλό, αλλά υπάρχουν κάποια στοιχεία ε, που μας δημιουργούν πρόβλημα. Θα κάνουμε και κάποιες τροπολογίες για τα NSA, τροπολογία 8 και για τις υποστηρικτικές υπηρεσίες υπάρχουν θέματα. Τα έχει φαντάζομαι υπόψη της Κομισιόν. Για τα φάψω όμως, ίσως εδώ διαφωνώ, γιατί ανησυχώ με κάποιες από τις τροπολογίες Μαρινέσκου. Γνωρίζω ότι η έκθεση είναι δύσκολη, όμως έχουμε κάποιες ανησυχίες. Και κάποια αλλαγή, κάποια μετονομασία πραγμάτων που δεν ε, μας ικανοποιεί και η άποψή του για τα φάψε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και ήμασταν ίσως οι μόνοι ξεκινήσαμε από κάτω προς τα πάνω. Κάποιες άλλες χώρες λένε να πάμε ανάποδα. Ε, αλλά πού σταματάμε, πού αρχίζουμε. Θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες από τα κράτη-μέλη που δεν βλέπω ότι εστιάζουν επαρκώ στο θέμα αυτό, γιατί πραγματικά όλοι μπορούμε να βγούμε κερδισμένοι σε όλα αυτά τα πράγματα. Ε, βλέπουμε λοιπόν τις τροπολογίες, τις μελετούμε και ευχαριστούμε τον κύριο Μαρινέσο και τη σκληρή του δουλειά. Περνάω στον κύριο Σασόλη που πάρα πολύ ευγενικά είναι εδώ σήμερα. Μια άλλη έκθεση λοιπόν που έχει μεγάλη σχέση με όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Και νομίζω θα πρέπει να τροποποιηθεί γιατί υπάρχει όπως είπα αυτή η ε, διασυνδεστώση ότι αφορά το όνομα. Είναι μια, ε, ένας οργανισμός ε, ασφάλειας, αλλά το να αρχίζουμε να παίζουμε με το όνομα και να αλλάζουμε ονόματα δεν νομίζω ότι έχει κάποιο νόημα εγχείρημα. Σε ό,τι αφορά τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο, υπάρχουν πολλοί, νομίζω 30 μέλη. Το να γίνουν 5 όμως, η Κομισιόν, ένας εκπρόσωπος και άλλοι 4, δεν είναι καλό αυτό. Δεν θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση. Ε, δεν θα έπρεπε να υπάρχει και κάποιος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν λέω ότι θα πρέπει να έχει συγκεκριμένο αριθμό μελών το διοικητικό, αλλά θα πρέπει να φαίνεται η εμπειρία ε, να εκπροσωπείται η εμπειρία και η τεχνική γνώση. Πέντε άτομα μόνο να επιφορτίζονται με τη λήψη αποφάσεων που θα επηρεάζουν πάρα πολύ ε, σημαντικά κομμάτια ε, που έχουν να κάνουν με τον εναέριο χώρο. Αυτό απλά σας το λέω. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Σασόλη λοιπόν θα καταθέσουμε κάποιες τροπολογίε, αλλά καταλήγοντας ε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο και για τις δύο εκθέσεις και να μιλήσω για τη χρήση των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Συνέχεια ανακύπτει αυτό και υπάρχουν κάποιες υποθέσεις ε, και κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να είναι κατάλληλες και ενδεδειγμένες αυτές οι κατεξουσιοδότηση πράξεις. Υπάρχουν όμως ε, πολλά άλλα μέρη και τομείς που δεν είναι κατάλληλες κατά την άποψή μου. Έξω και υπάρχουν και εκτελεστικές πράξεις που μπορεί ε, η Κομισιόν να μην θεωρεί ότι είναι ε, σωστό να τα ε, υιοθετεί. Αλλά πώς θα αφήσουμε χωρίς έλεγχο τα πράγματα. Δεν θα πρέπει να δούμε τι κάνουν και τα κρατημέλη. Σας αφήνω με αυτές τις σκέψεις ευχαριστώντας τους δύο εισηγητές και θα καταθέσω όπως είπα τροπολογίες. Ελπίζοντας να γίνουν δεκτές και ελπίζω αυτά τα δύο θέματα να δεκπερωθούν λίγο ταχύτερα από ό,τι στο παρελθόν ευχαριστώ. Το λόγο κύριο Αλχαντράουι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα και εγώ για να συμπληρώσω αυτά τα οποία είπαν οι προλαλήσαντες συναδελφοί μου. Καταρχάς, υπάρχει ένα πρόβλημα εκτέλεσης της νομοθεσίας. Αυτό είναι σαφές. Και πολλές φορές το έχουμε πει. Η νομοθεσία ναι μεν έχει ψηφιστεί, επιτόπου όμως δεν κινούνται τα πράγματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει γίνει και τίποτε. Αλλά πρόοδο δεν υπάρχει. Τουλάχιστον σε επαρκέ επίπεδο και φαίνεται να υπάρχει και ένα πρόβλημα εμπιστοσύνη. Συνάπτουμε συμφωνίε με τα κράτη-μέλη τελικά. και αν δεν έχουμε συγκεκριμένες κινήσεις εκ μέρους τους, δημιουργούνται προβλήματα σε ό,τι αφορά αυτά τα φάψη ιδίω. Επίσης, τι γίνεται με τα πιο σημαντικά κατόφλια, με τις πιο σημαντικέ ορικέ τιμέ, και τι γίνεται και με τα εμπόδια που υπάρχουν και τα οποία οδηγούν τελικά σε καχυποψία σε σχέση με τις οργανώσεις ελέγχου τη ενέργειας κυκλοφορία. Κατ' εμέ δύο είναι τα πολύ βασικά. Πρώτον, ό,τι έχει να κάνει με την κατανομή των εσόδων από τον αεροέλεγχο. Διότι αν θέλουμε να είναι πιο αποτελεσματικές οι διαδρομές, οι μετακινήσεις, τα δρομολόγια, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα έσοδα των ε, ενώσεων και των οργανώσεων που θα τροποποιηθούν. Και υπάρχει καχυποψία όσο δεν βρίσκεται λύση στο σημαντικό αυτό πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν ΚΑΤΕΜΕ να εστιάσει σε αυτό το θέμα και να διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί αυτή η καχυποψία δεν επιτρέπει και τη συνεργασία με αυτές τις οργανώσεις και δεν έχουμε πρόοδο. Δεύτερο, Δεν θα πρέπει και οι εργαζόμενοι να είναι με το μέρος μας, γιατί βλέπουμε καχυποψία και από την πλευρά των εργαζομένων του κλάδου, που δεν γνωρίζουν ακριβώς σε ποια κατεύθυνση οδεύουμε και ποιος είναι ο αντίκτυπος στην προσωπική τους περίπτωση στον καθένα. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να είναι πιο προβλεπτική στη δράση της Κομισιόν, proactive όπως το λέμε στα αγγλικά, να εξετάσει τις λύσεις τις πιθανές. Και σίγουρα πρέπει να υπάρξει καλή ε, θέληση. Και αυτή την καλή θέληση πρέπει να την καλλιεργήσουμε στον κλάδο. Ολοκληρώνοντας, σε ό,τι αφορά τις προτάσεις αυτές καθευτές κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι περιέχουν καλά στοιχεία και λιγότερο καλά στοιχεία. Σε ό,τι αφορά την αποσύνδεση, το decoupling αυτό, ε, έχω κάποια ερωτηματικά. Και με τις προστρικτικές υπηρεσίες δεν ξέρω, καλές φαίνονται, αλλά υπάρχουν νομίζω κάποια κάποιες υπερβολές προτάσεις της Κομισιόν. Αυτή από σύζευξη θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα σε τομεί που λειτουργούν καλά μέχρι τώρα. Θα μπορούσε να δημιουργήσει πρακτικά προβλήματα, δυσαρέσκεια. Όλα αυτά θα τα μελετήσουμε. Πρέπει να τα μελετήσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σύντομα. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Αλκαντράου και κυρίως με το τελευταίο σημείο που ανέφερε. Υπάρχουν προβλήματα σε αυτή την, ε, σε αυτή την πολύ μοδάτη, λέει ο πρόεδρος λέξη, το unbundling που το, το, το έχει κάνει καραμέλα η Κομισιόν, unbundling από εδώ, unbundling από εκεί, ε, και στις μεταφορές ε, κάθε είδους, εν πάση περιπτώσει. Και εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω πού τραβάει κανείς ε, τη διαχωριστική γραμμή από το κρίσιμο, μη κρίσιμο, ε, συστήματα προσγείωσης ας πούμε, ε, εκεί ειδικά σε περιπτώσεις κακού καιρού, τι γίνεται, θα κάνουμε unbundling και σε αυτό, μας απασχολεί. Δεύτερο, αυτό το οποίο ανέφερε και ο κύριος Δανέλης και ο κύριος ε, Αλκαντράουι προηγουμένως. Ο κύριος Αλκαντράουι, ο οποίος είναι όμως και παλιός διπλωμάτης, το έθεσε πιο διπλωματικά το θέμα. Εγώ θα ε, ε, έλεγα όχι μελήματα, όχι ανησυχίες, αλλά πραγματικά εναντίωση νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε το ζήτημα με μεγάλη, ε, με, κατεπίγουσα διαδικασία. Ξέρουμε ότι όταν υπάρχει έτσι μία μια πρώτη αντίθετη άποψη ευλάς προσωπικού μετά θα έχουμε οπωσδήποτε και κάποιες ε, άλλες συγκεκριμένες δράσεις ε, και τελικά θα καταλήξουμε με κλειστά αεροδρόμια, ε, με ε, πολύ άσχημη ψυχολογία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. Επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να αναλυφθεί άμεση ε, δράση όσον αφορά τις επαφές με όλους και το τονίζω όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κυρίως όμως με τους εργαζόμενους σχετικά με το ε, ΕΑΣΑ. Ε, τι να σας πω, δεν ξέρω εάν ε, στο νέο ρόλο της ΕΑΣΑ είναι σημαντικό να αναφέρεται και η ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αλλάζουν τα ονόματα. Εν πάση περιπτώσει, οι αλλαγέ όμω ε, σε αυτό το εκτελεστικό συμβούλιο ή διοικητικό συμβούλιο, αυτό είναι, είναι σημαντικό. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι θα ε, γίνει μάχη ε, για, τους, για τα μέλη της εκτελεστικής αυτής επιτροπής, εκτελεστικού συμβουλίου κτλ. Ε, σε αυτή την περίπτωση και αν ξεκινήσει έτσι μεγάλη μάχη, ίσως ε, θα έπρεπε ε, να παραχωρήσουν τη θέση τους οι Βρετανοί, ίσως στη Γαλλία, αν έχουμε Γάλλους και Γερμανούς σε αυτό το Συμβούλιο, ενδεχομένως τα πράγματα να λειτουργήσουν διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει όλοι να καθίσουν γύρω από το τραπέζι και κυρίως, το τονίζω, κυρίως να είναι υπόλογοι όλοι για τις ε, αποφάσεις ε, τις οποίες ε, παίρνουν. Γιατί διαφορετικά θα λέμε όλοι «Α, αυτοί οι βρωμογερμανοί φταίνε» ή «Αυτοί οι βρωμογάλοι» ή «Αυτοί οι κακοί Άγγλοι είναι αυτοί που φταίνε για την απόφαση». Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί οι επιπτώσεις ε, της σύνθεσης ε, του ε, Συμβουλίου μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικές και εάν ξεχωρίσουμε, διαχωρίσουμε πλήρως το ποιος αποφασίζει γιατί, τότε ενδεχομένως διατρέχουμε τον κίνδυνο να μην είναι κανείς υπεύθυνο για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Ο κύριος Μόλντουιν από την Κομισιόν. Καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω πάρα πολύ την, ε, Κομισιό, την Επιτροπή σας συγγνώμη, ε, για την πολύ ισχυρή θέση και στάση που παίρνει πάντα όσον αφορά τον ενιαίο ουρανό. Ε, και εμείς θέλουμε να πάμε πιο γρήγορα και εσείς μας πιέζετε διαρκώς και χαιρόμαστε γι' αυτό. Έχουν υποβληθεί και από τους δύο εισηγητές επικοδομητικές τροπολογίες, γι' αυτό λοιπόν θα είμαι σύντομος κύριε Προεδρή, σχετικά σύντομος. Όσον αφορά τα σχόλια του κυρίου Σασόλη, να τον ευχαριστήσω για την πολύ επικοδομητική του στάση. Οι προτάσεις, ε, του είναι ε, ε σωστές. Ε, τώρα, όσον αφορά αυτή την ιδέα που μας έχει υποβάλει για τον διαχωρισμό προσωπικού, είναι πολύ καλό επίσης ε, η δυνατότητα ε, των grants έτσι ώστε να γίνει πιο ευέλικτο το σύστημα εσόδων και αυτό μας ικανοποιεί ως πρόταση. Ε, κοιτάξτε, εμείς βαδίζουμε βάση της ε, κοινή ε, προσέγγισης, μας λέτε. Ναι, είναι γεγονός. Απ' την άλλη πλευρά είναι αλήθεια ότι σε αυτή την προσέγγιση καμιά φορά έχουμε και την αντίληψη το one size fits all. Αλλά γι' αυτό θέλουμε και τις απόψεις του Κοινοβουλίου και εν πάση περιπτώσει εμείς προσπαθούμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν προωθούμε διάφορες ιδέες. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η κυρία Φώστα όσον αφορά ε, της ε, κατεξουσιοδότηση πράξης. Έχουμε και μητροπολογία που σχετίζεται με αυτό. Εμείς ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε τα στάνταρ τα οποία είχαμε μέχρι τώρα και ε, νομίζω ότι τα όσα αναφέρονται στο άρθρο, ε, προβλέπονται στο άρθρο 290 της Συνθήκης Λειτουργίας μας ε, οδηγούν. Δεν θέλω να μειώσω την σημασία του ρόλου των, και της διαβούλευσης με τους εμπειρογνώμονες. Έχω την αίσθηση ότι εσείς έχετε μια τάση έτσι, να υποτιμάτε λίγο αυτήν την πρακτική. Πρόκειται όμως για μια στάνταρ πρακτική και δεν νομίζω ότι στην ουσία δημιουργεί οποιαδήποτε ε, διαφορετικά. Όσον αφορά, ε, διαφορά. Όσον αφορά τώρα το Συμβούλιο ή μάλλον τα Συμβούλια. Ε, αυτό ε, θα παίρνει τις ε, αποφάσεις για την ΕΑΣΑ με 32 μέλη. Θα αφορά τώρα το Executive Board, και αυτή είναι η κοινή απόφαση επίσης, είναι ότι προσπαθεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της, του οργανισμού. Θέλει να βοηθήσει στην ουσία λοιπόν την λειτουργία του οργανισμού. Ε, όταν τα κράτη-μέλη ε, θα έχουν δει στη λειτουργία του το πράγμα, ε, δεν θα είναι αρνητικά προσκύμενα προς την διαδικασία αυτή, γιατί στην ουσία όντως θα υπάρχει μια ανακύκληση των μελών. Όσον αφορά τώρα τον ίδιο τον οργανισμό πολλά ενδιαφέροντα σχόλια ακούσαμε. Συμφωνούμε απολύτως ότι η πρώτη δουλειά του οργανισμού θα είναι η ασφάλεια. Άλλωστε στο άρθρο 2.1 του κανονισμού αυτό υπογραμμίζεται με τεπιτάσεως. Αλλά θα υπάρχουν και άλλες ε, διαδικασίες οι οποίες ε, είναι πλέον ε, και πολύ της μόδας ας το πούμε. Δηλαδή και το περιβάλλον και όλες οι υπηρεσίες αεροναυτιλίας ATM ε, νομίζουμε ότι και ε, σε αυτούς τους τομείς μπορεί να αναπτύξει δράση ο οργανισμός, γιατί είναι δικιά του δουλειά. Ο κύριος ε, Σασόλη αναφέρθηκε στο θέμα της ασφάλειας και κοιτάξτε, δεν αλλάζει η ασφάλεια εάν αλλάξει το όνομα και αν δεν υπάρχει στον τίτλο δηλαδή η θέση, η αναφορά στην ε, ασφάλεια. Ε, νομίζω ότι ούτως ή άλλως ο ρόλος του ίδιου του οργανισμού και οι αποφάσεις που θα πρέπει να λαμβάνει και στο μέλλον θα είναι όλο και πιο ε, σημαντικές. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ για, τις, για τα σχόλια τα οποία ε, ε, μας έκανε ο κύριος Σασόλιος. Όσον αφορά τα σχόλια του κύριου Μαρινέσκου, δεν έχουμε πρόβλημα με τις περισσότερες τροπολογίες. Είναι λογικές. Ίσως θα ήθελε ο κύριος Μαρινέσκου να είμαστε πιο φιλόδοξοι, να έχουμε πάει παραπέρα αλλά ξέρετε καμιά φορά ε, υπάρχει ε, η μέθοδος η οποία δεν είναι πάρα πολύ εύκολη ε, πάντα να εφαρμοστεί όσον αφορά τους ορισμούς. Ναι, τροπολογίες 14, 15, 16 και 18 επ' αυτόν νομίζω ότι θα πρέπει να ευθυγραμμιστούμε με την ορολογία της ΔΟΠΑ. Όχι, τώρα να ξαναγυρίσω όμως, γιατί να πω ότι θέλουμε να ευθυγραμμιστούμε με την ε, ΔΟΠΑ. Γιατί κοιτάξτε, όταν ε, το 2004 ε, εγκρίναμε τους ορισμούς αυτούς, τους τροποποιήσαμε ελαφρά, τους έχουμε χρησιμοποιήσει για 10 χρόνια περίπου τώρα και δεν νομίζω ότι μπορούμε τώρα να τους αλλάξουμε. Δηλαδή δεν θα είναι και νομικός ορθό το να αλλάξουμε τους ορισμούς γιατί οπωσδήποτε θα απορρεύσουν ε, νομικές ε, επιπτώσεις ε, κυρίως όσον αφορά τα αναφερόμενα στις τροπολογίες 14, 15, 16 και 18. Τροπολογία 27, ρόλος της ΕΑΣΑ σε σχέση με τις εθνικές αρχές, αυτή είναι μια νέα ιδέα νέα λειτουργία. Δεν θα αντιταχθούμε καταρχήν. Αναρωτιέμαι πάντως εάν θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη ε, τροπολογία στον βασικό κανονισμό της ε, ε, ΕΑΣΕ. Τροπολογία 65 αναφέρεται στον ρόλο της ΕΑΣΕ πάντα και εδώ καταλαβαίνουμε ποιο είναι το σκεπτικό κυρίως ε, αναφέρεται δηλαδή στον εποπτικό ρόλο της ΕΑΣΕ στις διασυνοριακές ε, ε, μεταφορές, αλλά φαίνεται ότι εδώ στο δρόμο έχει χαθεί η έννοια της mutual recognition, αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών που υπήρχε στην αρχική, στο αρχικό κείμενο και εμείς θέλουμε να ξαναμπεί η ιδέα αυτή στο κείμενο ο ρόλος της ΕΑΣΕ όσον αφορά την εποπτεία είναι πολύ σημαντικός κατά την άποψή μας. Ε, τροπολογία 26 την έθιξαν αρκετοί ε, ε αρκετοί ομιλητές. Ε, κοιτάξτε αυτό το unbundling. Πρέπει να σας πω ότι θα συμφωνήσω μαζί σας ε, γιατί πρέπει να βγει από το λεξικό, να διαγραφεί αυτή η λέξη. Δημιουργεί πολλά προβλήματα, εγείρει πολλές αμφιβολίες. Ε, για την τροπολογία 76, συγγνώμη, όχι 26, 76, νομίζω ότι μέσω της τροπολογίας ε, κατά κάποιο τρόπο δεν ε, προχωράει πολύ το κείμενο και σας εξηγώ. Εάν συνεχίσουμε με την κοινή παροχή, ε, ε, παροχή υπηρεσιών, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εισαχθούν νέες υπηρεσίες, στήριξης εσωτερικών υπηρεσιών κτλ. και εσωτερικών παρόχων. Θεωρούμε ότι για να δημιουργηθεί ο, πραγματικά ο ενιαίος ουρανός και να λειτουργήσει θα πρέπει να υπάρχει αυτή η κυρία αντιμετώπιση. Τώρα, εάν θέλετε να επιμείνετε με το 76, ίσως ε, θα μπορούσαμε ε, να κάνουμε μία, εμείς ε, μία πρόταση διατύπωσης, έτσι ώστε τουλάχιστον και η τροπολογία, έτσι όπως την υποβάλλεται, να γίνει πιο αποτελεσματική. With the view of choosing και τα λοιπά. Κάτι να πούμε ότι με τελικό σκοπό την διαφορετική επιλογή ε, κτλ. Θα το δούμε. Θα το δούμε πάντα όσον αφορά την κοινή παροχή υπηρεσιών. 95 για το ΣΕΖΑ. Πρέπει να σας πω ότι εμείς ε, ε, πρόσφατα εγκρίναμε και έναν εφαρμοστικό κανόνα επ' αυτού. Πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς ότι θα πρέπει να ενταχθεί το πλήρες πλαίσιο της ΣΕΖΑ και όχι μόνο της ΕΣΥΠ που είναι πιο συσταλτικό. Τέλος. 108 για τη διαγραφή. Μπορούμε να καταλάβουμε ε, την, ε, ε, την περίεργη διατύπωση, αλλά κοιτάξτε, εάν διαγράψουμε όλη τη φράση, τότε θα αλλάξει και η ισορροπία με την έννοια Ίσως ε, θα πρέπει να διατηρήσουμε τουλάχιστον το τμήμα που λέει πρόσβαση στους λογαριασμούς κτλ. Κοιτάξτε, είπα ότι θα πω λίγα, τελικά μπαίνω σε λεπτομέρειες. Το ένα όσον αφορά το ΦΑΠΣ. Το αναφέρατε κι εσείς ε, και κύριε Μάλης και ο κύριος Κράμερ ε, και ο κύριος Γκρός και η κυρία Φώστερα, όλοι σχεδόν. Συμφωνούμε απολύτως ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν το ΦΑΠΣ είναι απολύτως ε, ουσιώδους σημασίας. Ε, τους τελευταίους μήνες, ε, αν όχι χρόνια, ακούμε πολλές ανησυχίες της Επιτροπής σας όσον αφορά τα ΦΑΠΣΑ και νομίζω ότι καλό ήταν που μας πιέζετε γιατί πραγματικά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα για δράση αλλά να μην τα πετάξουμε όλα, όπως λέμε να πετάξουμε το νερό του μπάνιου και μαζί και το μωρό. Ας κρατήσουμε αυτά τα οποία είναι ε, καλά και τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ε, και εάν, συν, ε, εάν συντονίσουμε τη δικιά σας πολιτική πίεση με μια δικιά μας νομική πίεση νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι. Πρέπει να σας πω ότι πρόσφατα συναντηθήκαμε και τους επικεφαλείς των ΦΑΜΣ Κεντρικής Ευρώπης και, ε, αυτοί θέλουν να προχωρήσουν τα πράγματα. Όσον αφορά τον ε, Γεώργ, θα σας πω ότι είναι ζωντανός, είναι μια χαρά, τον είδα πρόσφατα, δεν τον έχουμε κλείσει σε κανένα ντουλάπι. Είναι πάρα πολύ καλά ο κύριος Γιαζεμπόφσκι και ε, χέρι άκρας υγείας. Ξέρετε ότι ε, ε, ε, ο ρόλος του ήταν να δημιουργήσει αυτά τα φάψη και αυτό κάνει. Και γνωρίζοντας τον άνθρωπο, ξέρετε ότι όπως βοήθησε και εσάς και εξακολουθεί να θέλει να σας βοηθήσει, βοηθάει και εμάς πάρα πολύ. Όσον αφορά τώρα τους εργαζόμενους, τις οργανώσεις εργαζομένων και ό,τι όνομα και αν δώσουμε ε, στα θέματα αυτά, οπωσδήποτε ε, θα είμαστε αφελείς ε, και ανόητοι μάλλον, εάν δεν τους λαμβάναμε υπόψη και αν δεν καταλαβαίναμε ότι ασκούν πίεση και εγώ θα πω απλώς πίεση, δεν θα πω ότι είναι επιθετική ή εχθρική όσον αφορά τις προτάσεις αυτές. Βεβαίως κατανοούμε ότι υπάρχει ε, μια ένταση ε, όσον αφορά τις ε, προτάσεις. Ξέρουμε ότι κινήσεις πολύ πιεστικές σαν αυτές του Ιουνίου και του Οκτωβρίου δεν βοηθούν. Αύριο θα έχουμε μία ε, συνάντηση, θα προσπαθήσουμε ε, να έρθουμε σε επαφή με, τους, ε, με τις οργανώσεις, με τους, τους NSPs, με τους εργαζόμενους όλους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια συλλογική συζήτηση είναι γεγονός ότι υπάρχει μία πίεση προς μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη, ε, καλύτερη αποτελεσματικότερη σχέση κόστους, ωφέλους, ε, αλλά ε, αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι να ξέρουμε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους τι τους ενδιαφέρει περισσότερο, μέχρι πού είναι διατεθειμένοι να πάνε, πού θα στυλώσουν τα πόδια τους κτλ. Αυτά. Ε, πρέπει να σας πω ότι και σαν τελικό συμπέρασμα ε, συμμεριζόμαστε πολλές κοινέ απόψεις. Ο κύριος Σασόλη, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για, τις, για την εργασία τους, τις παρατηρήσεις που έκαναν. Πολύ ενδιαφέρουσες σημαντικές παρατηρήσεις. Βεβαίως θα τις δουλέψουμε. Ε, και θα λάβουμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία αυτά ε, στα πλαίσια των τροπολογιών. Τώρα, να κάνω μερικές γενικές παρατηρήσεις. Εμείς θέλουμε οργανισμό ισχυρό. Θέλουμε ένα ενωσιακό σύστημα διακυβέρνησης, διότι πιστεύουμε ότι μία διακυβέρνηση ενωσιακού ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Οργανισμού ε, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ε, διευθετεί τις, ε, τις θέσεις των κρατών μελών έτσι ώστε να ενισχυθεί η δύναμη απόφασης που μπορεί να έχει μια ενωσιακή απόφαση και ένα ενωσιακό πνεύμα ας πούμε. Αλλά θα πρέπει να βρούμε τη σωστή δύναμη, ούτε υπερβολικά πολύ ούτε υπερβολικά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 ε, όσον αφορά τώρα την εργασία και με τον συνάδελφο Μαρινέσκου, δεν θέλω ε, να υπερβωτέ καμένα και να πατήσω στα δικά του τα χωράφια, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει κυρίως η ασφάλεια να μας ε, απασχολήσει. Όσον αφορά τα διοικητικά συμβούλια, δεν μας απασχολεί μας αυτό, δεν θέλουμε να το πειράξουμε. Εμείς αναφερόμαστε μονάχα στο εκτελεστικό συμβούλιο, όχι στο διοικητικό συμβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο θα ορίσει ένα εκτελεστικό συμβούλιο Συμβούλιο. Εμείς είχαμε προτείνει να είναι τετραμελές, αλλά μπορεί βεβαίως να είναι περισσότερα τα μέλη. Φυσικά είναι δύσκολο να, να εμφυσίσει κανείς ενωσιακό ε, πνεύμα σε έναν ε, οργανισμό ή συμβούλιο. Θα πρέπει να βρούμε την πλέον αποτελεσματική λύση αλλά να έχουμε σταθερό σημείο εκκίνησης, ε, το οποίο θα πρέπει να είναι ε, αυξημένο ενωσιακό πνεύμα. Και κάτι ακόμα. Με ευχαριστεί δεν θα συμφωνήσω απολύτως βέβαια με την Κομισιόν. Ε, μπορούμε να συζητήσουμε περαιτέρω στις επόμενες εβδομάδες το θέμα. Πάντως συμφωνώ με την κυρία Φώστερ και με τον πρόεδρο Μπράιαν. Ίσως κάτι δεν ε, έγινε απολύτως σαφές. Πρέπει να σας πω ότι εγώ ε, κινούμενος έτσι από κάποιο, συντονισ... Ε, ε, κάποιο συντηρητισμό θα ήθελα να υπάρχει η λέξη ασφάλεια. Κατά την άποψή μου η λέξη, ο όρος ασφάλεια θα πρέπει να παραμείνει έτσι ώστε να καθορίζει ένα πλαίσιο εντός του οποίου και οι 28 χώρες υφίστανται αυτόν τον όρο, δηλαδή είναι σε θέση να ε, είναι ενεργοί παίκτες, να συμβάλλουν ενεργά στην ασφάλεια. Γι' αυτό εγώ θα προτιμούσα να παραμείνει ο, ο τίτλος του οργανισμού με συμπεριλαμβανομένη και του όρου ασφάλεια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. Είμαι βέβαιος ότι τις επόμενες εβδομάδες θα κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φώστερ νομίζω θέλει το λόγο πολύ σύντομα. Ναι, πράγματι πολύ σύντομα σχόλιο για τη σύνθεση του ή των συμβουλίων πράγματι 32 για το κύριο, το κυρίο συμβούλιο, αλλά υπάρχει ήδη ένα σύστημα Νομίζω 10 ή 12 από τις μεγαλύτερες χώρες, γιατί δεν έχουν πόρους ε, οι άλλες οι μικρότερες χώρες, που ήδη εκεί έχουν λιγότερους, λιγότερους ανθρώπους, οι οποίοι ασχολούνται με πολλά από αυτά τα ζητήματα. Άρα θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με αυτή την εναλλαγή, αυτούς τους πέντε εκ περιτροπή. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι λογικό, γιατί πρέπει να υπάρχει συνέπεια. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Ίσως πρέπει να βάλουμε έναν όρο. Θα τα πείτε, λέει ο πρόεδρο για 10 mm. δευτερόλεπτα κάτι, κύριε Μπόλμουιν. Ναι, δεν θέλω να επανέλθω, αλλά για να μην υπάρχει σύγχυση. Αυτό το συμβούλιο που λέει η κυρία Φώστα, δεν θα το πιστέψετε, λέγεται FAPS. Και αυτό, τέλος πάντων, υπάρχουν αυτά που είπατε, ε, τα συμβούλια με 10 μέλη, μπορούμε να δούμε ε, τον αριθμό, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην πραγματικότητα ε, είναι να ενισχύσουμε αυτή την προπαρασκευαστική διαδικασία, να ενισχύσουμε το σύστημα, όχι να αποδυναμώσουμε το ρόλο των κρατών μελών που πιστεύουν ότι διαδραματίζουν και πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα συμβούλια. Η περιτροπή η αναλλαγή αυτή που λέτε πράγματι δεν χρειάζεται να γίνεται κάθε χρόνο, έχετε δίκιο, θα το δούμε ο πρόεδρος. Μήπως καθυστερήσει, αυτό με ανησυχεί, γιατί ενδεχομένω ενδεχομένως ασκηθούν πιέσεις ε, στα κράτη-μέλη για το ποιον θα βάλουν, σε ποιο συμβούλιο, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, λοιπόν, 26 Νοεμβρίου λίγη προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Η εξέτασή του θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου και θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Μεταφορών στις 30 Ιανουαρίου. 26 λοιπόν Νοεμβρίου λίγη προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Επόμενο σημείο Τη μέσης διάταξης είναι το σχέδιο έκθεσης της κυρίας Λίχτενμπέργκερ για στατιστικές σχετικά με μεταφράσει εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών. Εύα. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ είμαι, εδώ. Σχόλια εκτός μικροφώνου από τον Πρόεδρο. Το θέμα των στατιστικών ακούγεται πάντα κάπως στεγνό και μη ενδιαφέρον, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον προσδορισμό των πολιτικών επιλογών. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επαναλαμβάνει δυστυχώς για μας ακόμη για μια ε, ακόμη φορά μεγάλο αριθμό προτάσεων ε, εκτελεστικών. Αυτό που θεωρώ εγώ σημαντικό είναι η καταγραφή όχι μόνο των μεταφορών ε, φορτίων σε ιστορικές πρωτοσοδούς, αλλά και επιβατών. Έτσι λοιπόν μπορούμε να καταγράφουμε και τα φέρει και τις κρουαζιέρες που είναι όλο και πιο συχνές, διαρκώς διευρύνει το σχετικό κλάδος, ιδιαίτερα στο Δούναβι, είναι πολύ συνηθισμένο πια φαινόμενο οι κρουαζιέρες στο Δούναβι. Και επίσης το λέω αυτό γιατί θα πρέπει ούτως ή άλλως να μας απασχολήσει σε μεταγενέστερο χρονικό ε, στάδιο το θέμα αυτό με τη διάσταση των υποδομών και πολλών άλλων. Για τις υποδομές δε, που όλο και πιο μεγάλη σημασία θα παίρνουν πιστεύω, κεντρική σημασία είναι η διαλειτουργική τερματική σταθμή, γέφυρες, ε, χώροι μεταπιβίβασης. Πρέπει δηλαδή να γνωρίζουμε πού πραγματικά, γι' αυτό χρειαζόμαστε στοιχεία, που πραγματικά υπάρχουν οι ανάγκες και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την φόρτωση από φορτηγά αυτοκίνητα αλλά και από σιδηροδρομικούς σταθμούς, διασύνδεση δηλαδή με σιδηροδρομικούς σταθμούς. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε και από εξοπλισμό και από διεύρυνση των υποδομών, ανάλογα δε και με τα καύσιμα που θα πρέπει να αξιοποιούνται. Όλα αυτά τα στοιχεία τα χρειαζόμαστε ώστε να γνωρίζουμε τι είδους τεχνικές προσαρμογές θα χρειαστούν. Υπάρχει δε ανάγκη να καταγράψουμε εάν εμφανίζεται η λεγόμενη τάση προς πιο καθαρά πλοία, cleaner ships, ή αν τελικά δεν έχει επαληθευτεί αυτή η πρόβλεψη. Και αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό με σοβαρότητα, θα επισημάνω ότι στο Κοινοβούλιο είχαμε κάνει μια ακρόαση πριν από λίγο καιρό, όπου συζητήσαμε και τις γραμμές στις πλωτές οδούς ε, ε, με την προοπτική της κλιματικής αλλαγής, το λιώσιμο των πάγων και παγετώνων και ενδεχόμενη επίδρασή τους στον υδάτινο ορίζοντα το του Δούναβη και άλλων ε, ποταμών διότι απολύπουσα στις ανασχετικής δράσης των παγετώνων υπάρχει κίνδυνος να επηρεαστεί σημαντικά το επίπεδο των υδάτων των ποταμών αυτών και θα πρέπει να το κοιτάξουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό θέλουμε στοιχεία στατιστικά που να μας επιτρέπουν να ρίξουμε μια ματιά υπεύθυνα στο μέλλον για το τι θα συμβεί. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Γκρός για τον κύριο Νταντά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια. Το κύριο Νταντά εκπροσωπώ εδώ, ζητώ συγγνώμη εκ μέρου του. Μας έχει επισημάνει στα ωραία του γαλλικά ότι συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με την εισηγήτρια την ευχαριστεί πολύ. Πρέπει να περιγράφονται και τα στοιχεία για τους επιβάτες. Εν γέννη πάντως διαρωτάτε εάν σε αυτές τις στατιστικές έρευνες κινδυνεύουμε να με αυτές τις στατιστικές έρευνες κινδυνεύουμε να επιβαρύνουμε υπερβολικά τον κλάδο ε, με γραφειοκρατικό επιπλέον φόρτο, γιατί θα πρέπει πάντα να διερευνάτε ποιο είναι υπεύθυνο, υπό ποιου όρου, πότε και πώ, για να διαθέσει τα απαιτούμενα στοιχεία. Και πρέπει να κοιτάμε τα στοιχεία να είναι χρήσιμα και όχι ε, οτιδήποτε μπορεί να διανοηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οτιδήποτε μπορεί να διανοηθεί κανεί να ζητήσει. Στόχοι σαφεί λοιπόν, αλλά με επισήμανση να αποφεύγονται οι διπλές, τριπλές, πολλαπλές αιτήσει για στοιχεία ή καταγραφές στοιχείων. Για δε την ε, επιτροπολογία και δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο έχει λόγο εδώ, πιο... θα πρέπει να έχει λόγο εδώ πιο ισχυρό, εδώ συμφωνεί με την εισηγήτρια ο εισηγητή και την ευχαριστεί και πάλι. Ο κύριος Αλκαντράου. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε. ουσιαστικά περνάμε στη νέα μέθοδο των κατεξουσιώδης και των εκτελεστικών πράξεων. Και πιστεύω ότι μπορούμε να διατυπώσουμε ε, κάποιες συστάσεις ε, όπως αυτές του συγητού και γι' αυτό και τις αποδέχομαι. Δεν χρειάζονται μόνο στατιστικές ε, για τη μεταφορά εμπορευμάτων αλλά και επιβατών και αυτό πρέπει να το ζητήσουμε από το Συμβούλιο. Αυτό είναι νομίζω σε αδρές γραμμές ε, αυτό που προτείνει η και μπορούμε να, ή η και μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Θέλουμε να υπάρχει ε, συνεκτικότητα των ε, στοιχείων. Και θα πρέπει σε ένα μεταγενέστερο στάδιο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα από τη χρήση αυτών των στοιχείων. Σε ό,τι αφορά το δικό μας μεταγενέστερο έργο θα μπορούσε να μας διευκολύνει στην Επιτροπή Μεταφορών κάτι τέτοιο. Θα στηρίξουμε λοιπόν τις προτινόμενες τροπολογίες. Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την εισηγήτρια Εύα Λιχτιμπέρκερ. Πιστεύουμε κι εμείς ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την προσαρμογή του κανονισμού στους όρους της συνθήκης Λισαβόνας για να τον βελτιώσουμε στο μέγιστο δυνατό, χωρίς βεβαίως να επιβαρύνουμε γραφειοκρατικά τις επιχειρήσεις, αλλά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε και ούτως ή άλλως έχουμε σε θέση μας κάποια από τα στοιχεία και πρέπει να καταγράφουμε ακόμη περισσότερα στοιχεία. Είναι κάτι πολύ καλό για να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα, η συλλειτουργικότητα, γιατί αυτό το επιδιώκουμε όλοι πιστεύω, να βελτιώσουμε την αξιοποίηση των διαφορών τρόπων μεταφοράς, αλλά ταυτόχρονα και για να βελτιώσουμε τους όρους μεταφοράς και όταν μιλούμε για τις ιστορικές πλωτές οδούς και όχι μόνο για φορτία αλλά και για ε, επιβάτες νομίζω ότι είναι πολύ καλή επιλογή να έχουμε τα στοιχεία αυτά για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε καλά. Ευχαριστώ κύριε Ενέσκου. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας καλημερίσω κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλου ιδιαίτερα στην εισηγήτρια, βέβαια, αλλά και όλα τα άλλα μέλη τη Επιτροπή σα για τα πολύτιμα σχόλια. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της αποσκοπούσε ουσιαστικά στην ευθυγράμμιση του εν λόγω κανονισμού προς τη συνθήκη της Λισαβόνας. Βέβαια, συμφωνούμε πλήρως με αυτά που είπατε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσει μέσω μιας μελέτης και με ένα πιο εναρμονισμένο τρόπο και τους πέντε τρόπους ε, μεταφοράς και τους σχετικούς κανονισμούς κάπως να τους ε, ευθυγραμμίσει, να τους ε, εναρμονίσει. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες για τη συλλογή δεδομένων, όπου ζητείται αύξηση των μεταβλητών, κατ' ουσίαν θα θέλαμε ως Κομισιόν προς το παρόν να εκφράσουμε με επιφύλαξη, διότι θα πρέπει να αναλύσουμε το αυξημένο βάρος και κόστος εκτός μικροφώνου σχολή της κυρίας Λίχτεμπέργκερ. Αυτά, ευχαριστώ. <laughs> Βεβαίω Εύα, να σχολιάσεις. Ναι, μόνο ένα σύντομο σχόλιο εδώ. Τα δεδομένα αυτά σε εθνικό επίπεδο είναι σχεδόν παντού υπαρκτά. Είναι δεδομένο αυτό. Και εδώ απλώς προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την καταγραφή τους κατά τρόπον ώστε να είναι συγκρίσιμα και ε, συμπιλήσιμα. Υπάρχουν ούτως ή άλλως ε, σε εθνικό επίπεδο τα δεδομένα αυτά. Δηλαδή δεν ζητούμε επιπλέον ε, επιβάρυνση των επιχειρήσεων. Αυτό που απαιτούμε είναι να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για να προγραμματίσουμε τις υποδομές της ενέργειας, Φερρυπίν. Δεν πρέπει να ξέρουμε πώς εξελίσσεται όλο αυτό το σύστημα. Ή θα πάμε στα τυφλά. Χρειαζόμαστε μια σαφή εικόνα ανάλογα με το τι θα συμβεί για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε. Για να έχουμε μια πιο καλή απεικόνηση της πραγματικότητας. Και αυτό μέσα σε ένα ε, τύπο, σε ένα format, το οποίο να μας επιτρέπει τα στοιχεία που προέρχονται από διαφορετικά κράτη να τα αξιοποιούμε ε, συλλογικά. Και πάντα όταν ε, κάνουμε κάποιες προτάσεις, Φερρυπίν, για τις υποδομές, προσπαθούμε να δούμε και άλλα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να έρθουν μπροστά μας σε λίγο καιρό. Ε, γι' αυτό κοιτάμε λίγο πιο μακριά και προσπαθούμε να συλλέξουμε στοιχεία στο δυνατόν πιο γενικά. Ευχαριστώ. 21 Νοεμβρίου λίγη προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών. Στην Επιτροπή Μεταφορών ψηφίζουμε στις 17 Δεκεμβρίου. Σας ευχαριστώ και περνάμε στο επόμενο θέμα που είναι ο κανονισμός ε, για τα στατιστικά στοιχεία για τις συνδρομικές μεταφορές όσον αφορά τις λογικέ στοιχείων για εμπορεύματα, επιβάτες και ατυχήματα. Μιχάλη Κράμερ. Ναι, δεν είναι εδώ διαφιλονικούμενο το θέμα και ευχαριστώ θερμά τους και οδησηγητές για την συνεργασία. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ και συγχαίρω τον Μάτσιο Εγκούς για την μεταφορά του 5% των ε, μεταφορών στις, ε, στους που προτείνει η Λευκή του Βίβλους και φυσικά εδώ θα χρειαστούμε για να προχωρήσουμε τις κατάλληλες στατιστικές. Εδώ υπόβαθρο της ε, έκθεσης είναι ο κανονισμός για την παραγωγή στατιστικών τσένων σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές και βέβαια και για, το, για τις υποδομές, την ενέργεια που χρειάζεται κτλ για να μπορούν να συλλέγονται λοιπόν καλύτερα στοιχεία, πιο γρήγορα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να είναι σχετικά εναρμονισμένος ο τρόπος με τον οποίο θα καταγράφω τα στοιχεία αυτά και πρέπει να, πρέπει να μην καταγράφονται πλέον τα ατυχήματα, διότι αυτά υπάγονται πλέον στην οδηγία ε, για τους σιδηροδρόμους, πάλι δική μου έκθεση στο παρελθόν, που καλύπτονται ε, και όσο του καλύπτονται από αυτήν. Υποστηρίζω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εισαγωγή απλοποιημένων κανόνων για τη δημιουργία στατιστικών τη Ένωση ε, σε μία έκθεση, δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλαπλέ εκθέσει. Προσαρμογή στον, ε, στη συνθήκη τη Λισαβόνα κατά πιο, ε, αυστη, με πιο αυστηρούς όρους. Δεν πρόκειται να σας αφήσουμε να μας φάτε τα κουλουράκια μας, είναι δικά μας και θα τα υπερασπιστούμε. Η Eurostat θα συνεχίσει την συλλογή των δεδομένων έχει ήδη καλή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Θα ήταν εσφαλμένο τόσο να τι αφαιρέσουμε τις ε, αρμοδιότητες, γιατί χρειάζονται, ε, χρειάζεται να διατηρήσουμε μια εικόνα της διαλειτουργικότητας. Συνεργασία λοιπόν καλύτερα και όχι μονομερής καταγραφή ή μονομερής δράση. Στο θέμα του, της συγχωρήπανσης και του της ε, τροχοπέδης, της σιωπηλή τροχοπέδης, με 80% της μεταφοράς των φορτίων από το σιδηροδρόμο, εάν εισαχθεί αυτή η τεχνολογία, ασφαλώς θα έχουμε μειώσει κατά 20% τουλάχιστον την στην Ευρώπη και βέβαια θέλουμε κάλυψη της υπερσυνοριακής διάστασης ώστε να αντιμετωπιστούν όπου υπάρχουν χάσματα στις ρυθμίσεις και να προβλέψουμε φερειπίν και τη μεταφορά ποδηλάτων μέσα της, ε, μέσω των τρένων. Και πρέπει να σας πω ότι 20 χρόνια μετά το τέλος ε, του σιδηρού παραπετάσματος ε, κλείνει ένα κενό 660 μέτρων, αγαπητέ Ματσιέ, στις ε, διασυνδέσεις δρομικέ μεταξύ Γερμανίας και Τσεχίας. Ε, αυτό νομίζω μπορούμε να το ε, πανηγυρίσουμε. Έχουμε καταφέρει κάτι το υπέροχο, κάτι το τεράστιο, κάτι το μοναδικό, 660 ολόκληρα μέτρα στους σιδηροδρομικούς ε, στις συνδρομικές διασυνδέσεις νομίζω ότι μπορούμε να σεμνηνόμεθα για το μεγάλο αυτό επίτευγμα και μας περιπτώσει 6 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα ή περισσότερα, ό,τι είναι, όπου υπάρχουν κενά και χάσματα θα πρέπει να τα καταγράφουμε για να τα προωθούμε και να τα καλύπτουμε εγκαίρως. Γιατί εκεί το θέμα δεν είναι οικονομικό τόσο. Επίσης ζητούμε απλούστευση των στοιχείων με, συμπληρωματική βέβαια τήρηση των προσδιαγραφών και στόχων της Λευκής Βίβλου. Αυτά ευχαριστώ και την Επιτροπή και τους συναδέλφους. Σε ευχαριστώ πολύ Μιχάλη για μια ακόμη φορά ε, και καλό θα ήταν να μπορούν να περνάνε τα τρένα από τα σύνορα για να χαροποιήσω και τους καλεσμένους από την SNCF. Είναι όνειρο για όλους μας όπως το όνειρο που είχε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, να περνάνε τα τρένα από τα σύνορα του χρόνου ίσως. Είπα ότι έχουμε από την SNCF πολύ νεαρούς, τουλάχιστον φαίνονται πολύ νεαροί. Είναι το μέλλον. Θέλω λοιπόν να φύγουν από εδώ έχοντας στο μυαλό τους ε, τα σχέδια να έρχονται, να φεύγουν, να περνάνε από τα σύνορα κτλ. Yeah, Freiburg and Στρασβούργο Κέλ. Μιλάμε για όνειρα θερινής νυχτός. Ο κύριο ε, Γκρός, πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα είπα, θέλα και εκ μέρου του σκιώδου συγητού του κυρίου Μπόρισοφ να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Κράμερ, για την πρότασή του. Ο κύριος Μπόρισοφ ιδιαίτερα επισημαίνει Πρώτον, την απέτηση να είναι αξιόπιστα τα δεδομένα που θα συλλέγονται. Φυσικά για τη διαδικασία έχει πολύ δίκαιο, Μίχελ, αλλά θέλουμε αξιόπιστα στοιχεία. Ε, δεύτερον, και αυτό το θίξαμε και στην άλλη έκθεση, να μην γίνεται επικάλυψη, να μην επαναλαμβάνει τη ίδια δουλειά, αλλά να είναι ε, συμπιλημένα και συμπιλήσιμα κατά το δυνατόν τα στοιχεία. Επαναλαμβάνω λοιπόν όχι επικαλύψεις, όχι επαναλήψη ε, έργου είναι κάτι το οποίο πάντοτε αναφέρουμε όταν ε, πρέπει σε δύο διαφορετικές κατηγορίες να καταγράφονται τα ίδια στατιστικά στοιχεία, χάνουμε χρόνο, κάνουμε περί δουλειά. Η ασφάλεια βεβαίως των υποδομών δεν μπορεί να λησμονηθεί και επίσης για να δώσω και μια δική μου παρατήρηση, είναι πολύ ενδιαφέρον και το θέμα αυτού του, αυτής της τροχοπέδης που ψιθυρίζει, όπως λέγεται στα γερμανικά. Αστείο μου φαίνεται λίγο, γιατί δεν υπάρχει βέβαια τροχοπέδι που να ψιθυρίζει, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είναι και λίγο πιο ήσυχο και μειώνει την ηχορύπανση, τόσο το καλύτερο. Αλλά όλα αυτά θα κρυθούν από την ποιότητα που θα εξασφαλίσουμε. Αυτές είναι οι τύχε που θέλω να υπογραμμίσω και ιδιαίτερα για τις μεγάλες χώρε που μερικέ φορέ λησμονούν και ότι έχουν κοινά σύνορα με μικρότερα κράτη και ω εκ τούτου δεν προβαίνουν σε απαιτούμενε ε, επενδύσεις. Θα ήταν καλό να ενισχύσουμε τις υποδομές, διότι δυστυχώς, δυστυχώς πολύ συχνά α, ελλείψεις στις υποδομές έχουν επίδραση και στην ασφάλεια και στην εισαγωγή περαιτέρω πιο σύγχρονων τεχνολογιών. Αυτά λοιπόν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η καταγραφή όλων αυτών των στοιχείων. Χαίρομαι. Η έκθεση αυτή μπορεί να ε, υποστηριχθεί από εμά πλήρω. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Κύριο Αλκαντράουι. Νομίζω τον κύριο Λιμπεράτσκι εκπροσωπείται. Είναι πράγματι αυτό είναι ο σκιώδη μα και δεν είναι πάνω σήμερα. Όμω μου είπε ότι τον ικανοποιεί πολύ ο τρόπος με τον οποίο συνεργάστηκε ο συγκεκριτής με τους κοιόδους συγκεκριτές και θεωρούν λοιπόν ότι λίγο πολύ μπορούμε να συμφωνήσουμε για όλα. Λίγο πολύ. Φυσικά είναι σημαντικές οι στατιστικές για τη δημιουργία μιας νέας πολιτικής, για να μπορούν να γίνονται συγκρίσεις, δικαιώματα επιδόσεων όπως είναι αυτό το επιβατοχιλιόμετρο ή το τόνο χιλιόμετρο βέβαια θα πρέπει να μπορούν να μετρώνται με τον ίδιο τρόπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό. Για μας ήταν σημαντικό να συμπεριλάβουμε και κάποια στοιχεία για να μπορούμε ε, να, μετα, να μετράμε δεν ξέρω αν το SIP κιλομίτες ε, αυτό ε, στις δημόσιες υπηρεσίες, σε συμβάσεις ε, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί για τα καθίσματα δηλαδή και αφού φαίνεται να το λαμβάνει ο εισηγητής υπόψη, συμφωνούμε και είμαστε άκρως ικανοποιημένοι. Άρα θα στηρίξουμε την πρόταση του εισηγητή. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και θα δούμε τι θα προκύψει. Κύριε Μάισνερ. Ναι, ευχαριστώ. Δεν εκπροσωπώ κανέναν αυτή τη φορά. Είμαι εγώ σκιώδης και ευχαριστώ τον εισηγητή κύριο Κράμερ για την έκθεσή του, για την καλή συνεργασία. Συμφωνούμε και εδώ σε μεγάλο βαθμό. Θέλουμε καταρχάς τα δεδομένα, αλλά ταυτόχρονα συμφωνούμε ότι πρέπει να επαναλαμβάνουμε δουλειά που γίνεται αλλού. Πρέπει να βελτιώσουμε την λειτουργία της όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει δηλαδή να μην περιπλέκονται τα πράγματα για τον σιδηρόδρομο και αφού υπάρχουν κάπου δεδομένα. Όχι βέβαια σε διαφορετικές κατηγορίες ή διαφορετικού τύπου δελτία, διαφορετικά χρώματα, όπως λέει ο κ. Γκρός, αλλά ε, ουσιαστικά στοιχεία να τα αξιοποιούμε. Βεβαίως θα πρέπει να καταγράφονται και τα βαγόνια που μεταφέρουν εμπορεύματα, αλλά και πού, πώς, από ποιον, ε, γίνεται η φόρτωση, μεταφόρτωση, εκφόρτωση. Αυτά όλα νομίζω ότι η Digimove Move τα έχει καλύψει, τα προβλέπει με το Recast. Γι' αυτό θέλουμε πάνω απ' όλα να εντοπίσουμε πού είναι το καλύτερο σημείο, η καλύτερη αρχή για την καταγραφή, ο καλύτερο φορέα για την συλλογή αυτών των καταγραφημένων στοιχείων, ώστε να τα αξιοποιήσουμε στο δυνατόν πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ, κυρία Ενέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα σχόλια και τις ε, τροπολογίες που προτείνετε. Διαβάσατε ότι στόχος της Κομισιόν ήταν να αναθεωρήσει και να απλουστεύσει τη συλλογή στοιχείων και βεβαίως να αποφύγει την επικάλυψη και διπλή καταγραφή πρέπει να πω ότι είχαμε πολύ καλή επαφή με την European Rail Agency και την ECR που, με την οποία υπογράψαμε υπόμνημα κατανόησης έτσι ώστε ε, να ξανα... αυτά τα, κατα, διπλά καταχωρισμένα να αναλαμβάνονται από αυτήν την, ε, την υπηρεσία. Ε, βεβαίως με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να αναλύσουμε σε βάθος ε, τα στοιχεία των δύο ε, πλευρών ε, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα μόνο καλό μπορεί να είναι. Επομένως, στόχος είναι ε, να ληφθούν τα στοιχεία αυτά από την Υπηρεσία Σιδηροδρόμων ε, και να κοινοποιηθούν μέσω της Eurostat. Ε, βεβαίως σημαντικός είναι και ο ρόλος που παίζει ο οργανισμός στην επιβεβαίωση της εγκυρότητας των στοιχείων αυτών. Ευχαριστώ. να, θα ήθελα να πω δύο λόγια ακόμα για κάποιες μεταβλητές ε, οι οποίες ε, είναι οι απαραίτητες, όντως θα πρέπει να δούμε με προσοχή έτσι ώστε να καταλάβουμε ποιες είναι οι στατιστικές πληροφορίες ε, και ποιες είναι οι πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως έχουν συλλεγεί από άλλες πηγές. Η πρόταση που έχετε ενώπιόν σας στην ουσία είναι απόφαση κοινή συμφωνίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών ε, και συζητήθηκε επί μακρόν σε τεχνικό επίπεδο στις αντίστοιχες ομάδες εργασίας στην Eurostat και βεβαίως είναι και αποτέλεσμα συμφωνίας με μεγάλους χρήστες των στοιχείων αυτών όπως ας πούμε η DigiMove. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μάικλ, θέλεις να πεις τίποτα. Ναι, και έχουμε Του τύπου από την Essence. Α, δεν είναι εδώ, φύγανε. Φράιμπουργκ Κόλμαρ. Αυτό, αυτή τη γέφυρα που γκρέμισαν στον προηγούμενο, στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τα γερμανικά στρατεύματα δεν μπορούμε να την ξαναχτίσουμε. Και θέλω να πω επίση ότι αυτή η γέφυρα, να, ύστερα από 70 χρόνια θα μπορούμε να πούμε να τα καταφέραμε, τη χτίσαμε. Α το κάνουμε λοιπόν τουλάχιστον αυτό αν ήταν εδώ αυτή η νεαροί της SNCF θα είχα να τους δώσω καθήκον να εκπληρώσουν έργο που δεν έχουν εκπληρώσει προηγούμενες τρεις γενναίες. Αλλά εμπάσχετος, τι καλά που θα ήταν, αυτό έχω να πω. για τους κοιόδης συγγητές, σου ευχαριστώ πολύ. Για την Επιτροπή σας ευχαριστώ πολύ. Για τη γραμματεία της Επιτροπής μας ευχαριστώ θερμά για την πολύ καλή συνεργασία και για τις... Ε, για τις σιωπηλέ ε, τροχοπέδες θα έλεγα, οι συστήματα παίδησης, όχι τα ψιθυρίζοντα συστήματα παίδησης, θα έλεγα ναι, είναι πολύ σημαντικό να καταγράφονται, έστω και ένα δευτερεύον θέμα, είναι απαραίτητο να έχουμε τις σχετικές γνώσεις. Και σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστώ. Προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών 21 Νοεμβρίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή 17 Δεκεμβρίου. Και τώρα παρακαλώ να πάμε και κλεισμένων των θυρών. Θα πετάξω στο διάδρομο όποιον δεν έχει εργασία και δει το Συμβούλιο, καταλαβαίνετε γιατί.